Okay. Good morning. Εντάξει, καλημέρα σας και πάλι. Να συνεχίσουμε τις εργασίες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ μετά την κοινή ψηφοφορία που είχαμε με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη από εκεί που την είχαμε αφήσει χθες το απόγευμα. Μετά τις μακροσκελέστατες πληροφορίε που είχαμε. Ακόμη δεν έχουμε δει το σημείο 37 με την επίβλεψη των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων. καθώς και τις λειτουργίες και επιχειρήσεις του Οργανισμού των Κρατών Μελών για την παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων. Ο κύριος Κοέλιου, ο εισηγητής, θα μας περιουσιάσει πώς έχουν τα πράγματα και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, ιδίως στον τελευταίο τριμερή διάλογο, που έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη. Α ακούσουμε το πώ έχουν τα πράγματα από τον εισηγητή μα τον κύριο Κοέλιο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ να σα ενημερώσω ότι ο προηγούμενο τριμερή διάλογο έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα μάλλον, την Τρίτη, και με τη βοήθεια των σκιωδών εισηγητών Κέλλερ, Βίξτρομ, Ένστ, Βαντόλφε και Κίρκοπ, καταλήξαμε σε μια τελική συμφωνία Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να ολοκληρωθεί η εξέταση του θέματος και να φτάσουμε σε μια συμφωνία προτού πριν λήξει η θητεία. Να τονίσω ότι τα δικά μας απαγορευτικά όρια ευτυχώς έγιναν σεβαστά. Πρώτον, ο κανονισμός αυτός αποτελεί μια σοβαρότατη βελτίωση σε σχέση με την ισχύουσα απόφαση. Σεβόμαστε τις αποφάσεις του δικαστηρίου για αντικατάσταση του κανονισμού αυτού εντό εύλογου χρονικού διαστήματο. Δεύτερον, από την αρχή εξηγούμε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγέ στο σύστημα και να βρεθούν αποκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προλάβουμε του θανάτους στη θάλασσα. Έπειτα υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες για την έρευνα και τη διάσωση ορίζονται οι περιπτώσεις κατεπηγωσών παρεμβάσεων και η υποχρέωση να αναλάβει κανείς δράση και να σώσει ζωές. Ακόμη και όταν βρισκόμαστε στο πλαίσιο της εποπτείας των ε, θαλάσσιων συνόρων, κάτι που είναι η νομική μας βάση, χρειάζεται να έχουμε συγκεκριμένους κανόνες ώστε να διοργανώνονται επιχειρήσεις ε, έρευνας και διάσωσης. Όμως μιλάμε μόνο για επιχειρήσεις που συντονίζονται από τη Frontex. Τέσσερα, έχουμε υποχρεωτικά μέτρα εντοπισμού σε περιπτώσεις συλλήψεων και τα μέτρα δίωξης είναι μόνο προαιρετικά. Ακολουθούμε έτσι το αίτημα του Κοινοβουλίου να υπάρξει διάκριση προκειμένου να δημιουργηθεί μία ιεραρχία βάσει της οποίας πάντοτε κατά πρώτον θα υπάρχει εντοπισμός προτού υπάρξουν μέτρα καταστολής. Και πέμπτον, έχουμε διαγράψει την δυνατότητα επαναπροώθησης μέσω της θάλασσας. Υπάρχει η δυνατότητα προειδοποίησης ή διαταγής προς το σκάφος, να μην μπει στα χωρικά ύδατα, αλλά όχι κάτι άλλο. Έξι. Ε, προβλέπουμε την ανάγκη να επιδειχθεί μεγαλύτερη αλληλεγγύα. Βασιζόμαστε στην αρχή της αλληλεγγύης. Η κατανομή της ευθύνης και η αλληλεγγύη είναι ένα απαραίτητο παράγοντα για να βεβαιωθούμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών των ατόμων γίνονται πλήρως σεβαστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο, θα πρέπει να επιβάλλουμε την αρχή τη μία επαναπρόθεση. Έχουμε μη επαναπροθεση Έχουμε ένα πολύ ισχυρο, μια πολύ ισχυρή ιδεολογική σκέψη, η οποία καταστά σαφέ, αναφέρεται μάλλον με σαφήνεια στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και έχουμε και το άρθρο 4, όπου έχουμε προβλέψει πολλές βελτιώσεις. Το δικαίωμα στη ζωή, ο σεβασμός της αρχής της μη επαναπροώθησης είναι στην καρδιά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, που πρέπει να βεβαιωθούν για την πλήρη υλοποίησή τους και το σεβασμό τους. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία της, καθώς και τη Λιθουανική και Ελληνική Προεδρία. Νομίζω όλοι εργαστήκαμε σκληρά, προκειμένου να βρούμε μία λύση πριν τις εκλογές. Εάν και τα δύο θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, επιβεβαιώσουν ότι συμφωνούν με το κείμενο στο οποίο καταλήξαμε ως συμφωνία στον τριμερή διάλογο, θα καταλήξουμε και θα πετύχουμε να αντικαταστήσουμε την απόφαση του Συμβουλίου στο δυνατόν συντομότερα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο. Δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο. Όχι, ο κύριος Μπρόγκς. Θέλετε το λόγο πριν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Προεδρία. Θέλετε να παρατηρήσετε κάτι. Η αρχή της με επαναπροώθησης αναφέρθηκε και πάλι. Μιλάμε για μια ελευκό επιταγή, για έναν άγνωστο αριθμό ανθρώπων που έρχονται από διάφορες χώρες αυτό στην ουσία σημαίνει ότι οποιοδήποτε φτάνει στην Ευρώπη και από μια επικίνδυνη χώρα ενδεχομένω δεν μπορεί να επιστραφεί στη χώρα του. Εάν καταλήξουμε λοιπόν στο λογικό ή παράλογο συμπέρασμα, είναι ότι επιτρέπουμε στους πληθυσμούς των χωρών αυτών να μείνουν στα εδάφη μας. Εάς φέρουμε όλους τους πληθυσμούς των επικίνδυνων χωρών στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ας φερουμε ολους τους πληθυσμους των επικινδυνων χωρων στην ευρωπη ευχαριστουμε κυρια σαρχεντινη Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εισηγήτριά μας ήταν η κυρία Σκά Κέλλερ, αλλά δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Ενημερώθηκα όμως για την τελευταία συνεδρία των σχεδόν από την ίδια και οι πράσινοι πραγματικά θέλουν να ευχαριστήσουν τον Κάρλο Κουέλιου για, το, για την πολύ καλή του δουλειά Πραγματικά πιστεύουμε ότι η διατύπωση που χρησιμοποίησατε είναι πολύ ε, ισχυρή και κατανοητή για τη μία επαναπρόθεση και ευτυχώς, έστω και τελευταία στιγμή, υπάρχει ε, κάτι για την νομική αρρωγή που πρέπει να προσφέρεται στους ανθρώπους ακόμα και αυτούς που βρίσκονται σε σκάφη. Βεβαίως ο μεγάλος μας αγώνας παραμένει ότι η απόφαση αυτή επιτρέπει τον αποβασμό των ανθρώπων σε τρίτη χώρα. Το αν αυτό θα γίνει μόνο θεωρητικός ή θα υλοποιείται και στο μέλλον είναι κάτι που απομένει να το δούμε. Όμως πραγματικά δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που τα κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο να πετάξουν κατά κάποιο τρόπο τους πρόσφυγες σε τρίτες χώρες. Φαντάζομαι ότι τότε θα πρέπει να προσφύγουμε είτε στο Στρασβούργο είτε στο Λουξεμβούργο σε ένα από τα δικαστήρια διότι ακόμη και αν έχετε προβλέψει κανόνες και χέγγια που τα βρίσκουμε πολύ καλά και ακόμη και αν ισχύσουν, παρόλα αυτά κάποιοι δεν θα μπορούν να ε, ε, τυφούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα που αποσπάσατε. Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς? Όχι. Ας ακούσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Προεδρίας. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Χίλη. Η κυρία Χίλη. Κυρία Χίλη. Καλημέρα σας και ευχαριστώ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και το Κοινοβούλιο καθώς και την Προεδρία για την πρόοδο που επιτύχαμε στο θέμα αυτό. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα διότι θεωρούμε ότι το κείμενο, το συμβαστικό κείμενο επιτυγχάνει τους περισσότερους από τους στόχους του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ και ελπίζουμε το συμβαστικό αυτό κείμενο να επιβεβαιωθεί από τους δύο συνομοθέτες. Ωραία. Και από την Ελληνική Προεδρία, κύριο κ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους τους εισηγητέ και όλε τις πολιτικές ομάδες διότι συνέβαλαν με την επικοδομητική του τάση στο να πετύχουμε έναν συμβιβασμό. Νομίζω η ισορροπία που εξέφαμε είναι σωστή ως αποτέλεσμα του τέταρτου άτυπου τριμερούς διαλόγου. Αυτό ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και καταφέραμε να σεβαστούμε τις ε, περιοριστικές ε, διορίες και προθεσμίες που είχαμε στα χέρια μας, ώστε να έχουμε ένα νομοθετικό κείμενο πριν από τις ευρωεκλογέ. Το κείμενο είναι ισορροπό, προβλέπει τα σωστά δικαιώματα για τους ανθρώπους ε, με το σωστό πεδίο, καθώς και καλεί τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τους σωστούς κανόνες και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις της Frontex. Ευχαριστούμε για το τελικό αποτέλεσμα και ελπίζω από την πλευρά της Προεδρίας να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα αυτό στην Κορεπέρ σήμερα από την πλευρά του Συμβουλίου και από την πλευρά του Κοινοβουλίου στις 20 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή Λίμπε. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Κολέτσι. Δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις για την παρουσίαση αυτού του τριμερούς διαλόγου το θέμα του κυρίου Κοέλιου. Κύριε Κοέλιο, έχετε για τελευταία φορά το λόγο, αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση. Ναι, απλώ να ε, απαντήσω στην κυρία Σαρχεντίνη. Ευχαριστώ για την ε, συνεργασία σα και τη βοήθειά σα σε αυτό το φάκελο. Όλη τη στήριξη των πρασίνων, ιδίω για σημαντικέ τροπολογίε όπω οι 7 που διατηρήθηκαν στο κείμενο. Να πω ότι κατά την άποψή μου δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τον αποβασμό σε τρίτε χώρε, αλλά μπορούμε να προβλέψουμε χειροπιαστούς κανόνες. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Όπως γνωρίζει η κυρία Σαρχεντίνη, ως τώρα καμία επιχείρηση της Frontex δεν κατέληξε σε αποβασμό σε τρίτες χώρες. Δεν μιλάμε λοιπόν για κάτι που συμβαίνει συχνά. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί και ποτέ. Βεβαίως πρέπει να προβλεφθούν κανόνες ώστε να αποκλειστεί μια τέτοια δυνατότητα. αλλά νομίζω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να πετύχουμε συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο. Κλείσαμε και με αυτό το σημείο. Να σας ανακοινώσω ότι στις, ως τις, στις 10 μάλλον θα έχουμε εδώ την ε, διαμεσολαβήτρια ε, την Έμιλι Ορέλη και τον ε, διευθυντή του Frontex και θα έλεγα μέχρι να έρθουν οι προσκεκλημένοι μας να κάνουμε 5 λεπτά διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε 5 λεπτά για να την περιμένουμε. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.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 κάνετε κάποια ησυχία για να ξαναρχίσουμε. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Τέλος του διαλύματος. Έφτασαν οι προσκεκλημένοι μας στο Προεδρείο. Έχουμε την τιμή να υποδεχόμαστε την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, νέο εκλεφίσα, Ξέρουμε ότι ανέλαβε τη θητεία της γιατί ανανεώθηκε η θητεία του Ευρωπαίου Δημοσιολάβητη Η νέα Ευρωπαϊκή Δημοσιολάβητρια λοιπόν είναι η κυρία Έμιλι Ο Ράιλι. Ήδη από τον Μάρτιο του 2012 υπήρξε έκθεση για την Frontex και σύσταση τον Απρίλιο του 2013 ενώ ειδική έκθεση τον Νοέμβριο του 2013 όπου η Frontex απέρριψε μία από τις συστάσεις. Εδώ έχουμε την ε, κυρία Οράιλη λοιπόν για να μας παρουσιάσει την έρευνα για την ειδική έκθεση αυτή και μετά έχουμε τον κύριο Ιλκάινεν, Ιλκα Λάιτινεν μάλλον, που μας τιμά εδώ με την παρουσία του, τον διευθυντή του Frontex για να μας παρουσιάσει τη λειτουργία του οργανισμού που ξέρετε όλοι πολύ καλά πώς επηρεάζει και το δικό μας έργο. Και μετά θα έχουμε την κυρία Γιγκέγκορ και τον κύριο Κέσλερ που είναι συμπρόεδροι του Συμβουλευτικού Φόρουμ του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα της Frontex του Frontex που θα μας παρουσιάσουν τη γνωμοδότηση του Συμβουλευτικού Φόρουμ για τα θέματα αυτά. Η κυρία Ιγι δεν έχει φτάσει ακόμη, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε έχει βρεθεί παγιδευμένη σε κυκλοφορική συμφόρηση. Αλλά θα ακούσουμε τώρα την παρουσίαση της ειδικής έκθεσης από την κυρία Ωράιλη. Uh, uh, σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας ενημερώσω για την ειδική έκθεση που προετοίμασα σε σχέση με την ε, Frontex, τον οργανισμό ο οποίος ε, επικουρεί τα κράτη-μέλη στην επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων τους. Ο... Η έκθεσή μου αναφέρεται στο κατά πόσον γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει να πω ότι η συνεργασία μας κατά τη διάρκεια της έρευνας με την Frontex ήταν εξαιρετική και οι απαντήσεις που έλαβα στις 13 ε, από τις ερωτήσεις μου και στις στάσεις μου ήταν ε, ε, ικανοποιητικές. Ωστόσο, δεν έγινε δεκτό το έτοιμά μου να δημιουργηθεί ένα εσωτερικό σύστημα ελέγχου και γι' αυτό προετοίμασα την ειδική έκθεση. Δεν θεωρώ ότι ένα τέτοιο σύστημα θα επέλυε όλα τα προβλήματα, αλλά θα ήταν τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα έτσι ώστε να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως εκείνα ε, που ε, καθιερώνονται στη θεμελιώδη χάρτη ε, θεμελιωδών ελευθεριών και μας δεσμεύουν όλους. Η παράνομη μετανάστευση, η δημιουργεί μια μεγάλη πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει μια σύγκρουση των επιδιώξεων μεταξύ της προσπάθειας εξέτασης με νόμιμο τρόπο, με τρόπο σωστό των αιτήματων ασύλου και του ελέγχου των συνόρων. Και η Frontex βρίσκεται στην καρδιά αυτής της σύγκρουσης. Μέσω του κανονισμού που ζητά πλέον ε, ρητά από την Frontex να σέβεται την χάρτα ανθρωπινών ε, δικαιωμάτων και να παρακολουθεί κατά πόσο αυτά τα δικαιώματα γίνονται σεβαστά και από τα κράτη-μέλη στις κοινέ επιχειρήσεις. Έχει δημιουργηθεί ένας κώδικος που διέπει την ε, λειτουργία των επιχειρήσεων και τη δημιουργία επίσης ενός συμβουλευτικού συμβουλευτικού φόρουμ με την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτά είναι σημαντικά βήματα. Τον Μάρτιο του 2012 ξεκίνησε μια έρευνα από τον Σιολαβητή για να εξετάσει κατά πόσον η Frontex τηρεί τι δεσμεύσει που αναλαμβάνει από τη Χάρτα και τον σχετικό κανονισμό. Διαπιστώσαμε ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδο. Ωστόσο, Διαπιστώσαμε επίση ότι δεν είχε δημιουργηθεί ένα μηχανισμό εσωτερικό στην Frontex που να ελέγχει τι καταγγελίε για παραβιάσει. Και θεωρώ ότι αυτή, αυτό το γεγονό ότι δεν υπάρχει αυτό ο μηχανισμό είναι σημαντική έλλειψη στον τρόπο οργάνωση τη Frontex. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη καταγγελίε για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι επιχειρήσει. Επίση σημαίνει ότι όσοι καταγγέλουν τέτοια προβλήματα δεν έχουν δικαίωμα, δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν απάντηση αμέσω από τη Frontex κάτι το οποίο σημαίνει ότι καταγγελίε για παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, παραμένουν χωρί να δοθεί απάντηση σε αυτέ, χωρί να δοθεί συνέχεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλουν ότι ε, παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα του δικαιώματα στη διάρκεια των επιχειρήσεων τη Frontex. Και είναι λυπηρό το γεγονό ότι η Frontex δεν έχει δημιουργήσει αυτόν τον μηχανισμό. Αποτελεί. Ε, θεωρεί ότι αποτελεί αυτό αρμοδιότητα το κράτους μέλους στο οποίο έγινε η παραβίαση, στο οποίο καταγγέλλεται ότι έγινε η παραβίαση. Ωστόσο, αυτή η νοοτροπία, αυτή η λογική έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου η Frontex ρίχνει τη βάλα στα κρατημέλη και αντιστρόφως. Δεν θεωρώ ότι αυτή η λογική είναι σωστή. Όταν υπάρχει μια κοινή επιχείρηση στην οποία τα κρατημέλη συμμετέχουν με την, επιχειρούν από κοινού με τη Frontex και η Frontex έχει ευθύνη. Η ευθύνη προκύπτει από το γεγονός ότι η Frontex ε, δημιουργεί ε, τα πρότυπα, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στις κοινέ επιχειρήσεις που σχεδιάζει και είναι ακριβώς ο ευρωπαϊκός οργανισμός ο οποίος επιτήρει τα εξωτερικά σύνορα. Σε, κάθε περίπτωση έχει κρίσιμο ρόλο στην επιτήρηση των ε, σύνορων. Αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω και δέχομαι τον ισχυρισμό ότι λίγα από τα μέλη του προσωπικού της Frontex συμμετέχουν στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, δεν δέχομαι ότι οι αρμοδιότητες είναι τόσο ξεκαθαρισμένες και τόσο ξεκάθαρες μεταξύ των δύο φορέων. Πολύ συχνά ε, αυτές οι παραβιάσεις μπορεί να έχουν διαπραχθεί, καταγγέλλεται ότι, ε, ότι ε, διαπράχθηκαν από μέλη της Frontex που φέρουν στολή με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και είχαμε περιστατικά τραγικά πρόσφατα όλοι. Και δεν είναι σωστό να υπάρχει μια τόσο περίπλοκη, ένα περίπλοκο πλέγμα σχέσεων και να μην είναι ξεκάθαρο ποιος οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Οποιουσδήποτε έχει αρμοδιότητα και λειτουργεί ως εκπροσωπώντας ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να ε, λογοδοτεί ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ανάμεσα σε αυτά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ανθρωπιστικές καταστροφές που όλοι διαπιστώσαμε, που όλοι ε, είδαμε στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύουν πόσο η δράση της Frontex επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα εκείνων που επιδιώκουν προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πραγματοθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που ε, καθιερώνει η Χάρτα Ανθρωπινών ε, Δικαιωμάτων και Θεμελιδών Ελευθεριών, πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός εξέτασης των καταγγελιών. Η Frontex ε, ισχυρίζεται ότι δεν έχει τη νομική βάση για να δημιουργήσει έναν τέτοιον μηχανισμό. Αυτό που ζητάμε δεν, είναι, δεν, ζητάμε από τη Frontex να κάνει μια διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου ή να αντικαταστήσει την Επιτροπή στο ρόλο της ως θεματοφύλακα των συνθήκων. Αυτό που τη ζητάμε να κάνει είναι να εφαρμόσει την αρχή της χρηστής διοίκησης, την οποία οφείλει να ακολουθεί οποιαδήποτε ε, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχεται καταγγελίες, δηλαδή να απαντά στις καταγγελίες τις οποίες δέχεται. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank your... Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ας ακούσουμε τώρα τον ε, ε, επικεφαλής της Frontex, τον κύριο Lightning. Ας ακούσουμε την άποψη της ε, Frontex. Λοιπόν, από τον κύριο Λάιτινεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους και όλες. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για το γεγονός ότι οργανώσατε αυτό το γεγονός. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον ε, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Θα σας υπενθυμίσω. Σας υπενθυμίσω ορισμένα θέματα. Πρωτού έρθουμε στην ουσία αυτού του θέματος. Πρέπει να κρατήσουμε τρία πράγματα στο μυαλό μας για την ε, μετανάστευση, για την αντιμετώπιση του εγκλήματος, για τη διευκόνηση της ε, καλή πίστη μετακίνησης μεταξύ των συνόρων. Έχουμε, περί... Έχουμε περίπου 700, 700 ε, εκατομμύρια ε... περάσματα των συνόρων. Τρίτο στοιχείο που αφορά τις αρμοδιότητες και είναι κάτι το οποίο ε, το συζητάμε από το 2005 όσο θυμάμαι. Ποιος έχει την αρμοδιότητα, μάλλον η αρμοδιότητα για την επιτήρηση των συνόρων σύμφωνα με τις ε, συνθήκες είναι των κρατών μελών. Συγχρόνως όμως η Frontex επομίζεται τις δικές της ευθύνες και ορισμένε φορέ αυτέ οι ευθύνε είναι σαφώς καθορισμένες, γενικώ όμως ερμηνεύονται με διαφορετικούς τρόπους. Το επόμενο σημείο που θέλω να θίξω έχει να κάνει με την εφαρμογή του άρθρου 26α του κανονισμού της Frontex, όπως έχει τροποποιηθεί το 2011. Λέει το άρθρο αυτό ότι η Frontex θα θεσπίσει ένα αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης του Τη εφαρμογή του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλε τι δραστηριότητε τη. Σε ό,τι αφορά την ίδια την έρευνα, αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα, είναι ότι ήταν μια έρευνα η οποία ξεκίνησε με δική μας πρωτοβουλία και ήταν απόρρια της 13ης ε, σύστασης που ανέφερε προηγουμένως η διαμεσολαβήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε γενικά ικανοποίηση από την πλευρά της, του γραφείου του διαμεσολαβητή για την αντιμετώπιση από την πλευρά της ε, Frontex για τις 12 συστάσεις από τις συνολικές 13. Εδώ θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφές για το εξή σημείο. Η Frontex δεν αρνήθηκε καμία από τις συστάσεις που είναι η σύσταση υπαριθμών 13M που λέει θα πρέπει να λάβει όποιες ε, είναι απαραίτητες δράσεις για να αντιμετωπιστούν τα παράπονα σε όλες τις δραστηριότητες της Frontex που μπορεί να υποβληθούν από άτομα και τα οποία βρίσκονται στο δημόσιο συμφέρον και επίσης ζητείται από τη Frontex να δώσει την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Αυτή ήταν λοιπόν η σύσταση τη, της ε, διαμεσολαβήτριας η οποία οδήγησε στην απάντηση που δώσαμε εμείς προς το γραφείο του διαμεσολαβητή. Δεν αρνούμεθα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η σύσταση αλλά θέλω να κάνω μια παραπομπή στα καθήκοντα του υπεύθυνου για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν έχει καμία αρμοδιότητα στα πλαίσια δρασεών συντονισμένων με τα κράτη-μέλη ε, και τη Frontex. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ένας τρόπος για να αποσύσουμε τις ευθύνες μας. Είναι λοιπόν αυτή η 13η σύσταση, η σύσταση M για την οποία αναφερόμαστε. Το θέμα αυτό, όπως είδαμε, είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας. Όπως αναφέρθηκε και από τη Μεσολαβήτρια, ο κανονισμός της Frontex δεν μας δίνει σαφείς ρήτρες για τα θέματα αυτά και γίνεται το θέμα αυτό σε σχέση με την αρμοδιότητα των <clears throat> φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των κρατών μελών. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο παραμένει ασαφές και πρόκειται για τον όρο που αναφέρεται στην έκθεση προς το δημόσιο συμφέρον μέσα εισαγωγικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω. Να σας πω τώρα τι έχουμε ήδη και στη συνέχεια μπορούμε να δούμε τι ακόμα μπορεί να επιτευχθεί σε επίπεδο βελτίωσης. Έχουμε την εμπειρία να αντιμετωπίσουμε παράπονα. Υπάρχουν παράπονα τα οποία προκύπτουν από τους ε, αξιωματούχους της Frontex οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες από άτομα και από Μίκιο που εμπλέκονται. Έχουμε ήδη τρεις διαδικασίες που ισχύουν για αυτά. Ε, την διαδικασία για τα σοβαρά επεισόδια, τον κώδικα συμπεριφοράς που έχει συγκεκριμένες πρόνοιες και τις ε, μόνιμες ε, διαδικασίες, τις Standard Operating Procedures, SOP. Για το άρθρο 26α του κανονισμού της Frontex, το οποίο ζητά από τον φορέα αυτό της Frontex να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό μηχανισμό εποπτείας. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο υλοποίηση και την επόμενη εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο, θα, το Διαχειριστικό Συμβούλιο θα αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά και στη συνέχεια θα υπάρξει η έγκριση για τη δημιουργία αυτού του μηχανισμού. Επίσης το Συμβουλευτικό Φόρουμ, επειδή έχουμε τον, ε, ένα από τους συμπροέδρους του Συμβουλευτικού Φόρουμ εδώ παρόντα, ε, θα παίξει κάποιο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε πέντε συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα από τα πάγια θέματα στην ημέρηση διάταξη, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα συμβάντα αυτά, τα οποία έχουν και επίπτωση στα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχει λοιπόν τακτική συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών για τα θέματα αυτά σε κάθε μία από τι συναντήσει μα αυτέ πέντε φορέ το χρόνο. Αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό εδώ και στο οποίο αναφέρθηκε και η διαμεσολαβήτρια είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τι διάφορε κατηγορίε του προσωπικού οι οποίε εμπλέκονται σε δραστηριότητε τη Frontex. Εκεί που έχουμε τις περισσότερες δυνατότητε να επηρεάσουμε τα πράγματα είναι σε σχέση με το προσωπικό της Frontex. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες οι οποίοι εργάζονται για τη Frontex αλλά οι οποίοι ε, μισθοδοτούνται από τα κράτη-μέλη. Η τρίτη κατηγορία είναι μια νέα κατηγορία η οποία έχει θεσπιστεί από το νέο κανονισμό της Frontex. Είναι οι λεγόμενοι προσκεκλημένοι αποσπασμένοι αξιωματούχοι και υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για το δικό τους ρόλο. Αυτά είναι τα άτομα που έχουν το καθήκον της στήρισης της ε, νομοθεσίας κατά τη διάρκεια των ενεργειών της Frontex. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που έχουν βάση εξουσιοδότησης εξουσίας είναι η τρίτη αυτή κατηγορία. Οι προσκεκλημένοι αποσπασμένοι αξιωματούχοι των κρατών μελών οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Έχουμε επίσης και κάποιες άλλες κατηγορίες όπως είναι οι διερμηνείς κτλ. Έχουμε λοιπόν ένα είδος τριγώνου όπου πρέπει να δούμε όλες τις δυνατότητες για να επηρεάσουμε την συνολική διαδικασία. Όσο πιο πολύ προχωρούμε προς την κατεύθυνση των κρατών μελών, όσο λιγότερη δυνατότητα ε, παρέμβασης έχουμε εμείς και τόσο περισσότερο τα κράτη-μέλη αποφασίζουν περί του πρακτέου. Αυτό είναι λοιπόν ένα από τα ουσιαστικά σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη εδώ. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν στη συνέχεια. Αν συνοψίσω, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε τους κανόνες, έχουμε τα πρότυπα, έχουμε τις απαιτήσει και έχουμε την ανάγκη να αναπτύξουμε περαιτέρω τις πρακτικές μας. Ξεκινώντας από το σύστημα παρακολούθησης και αναπτύσσοντάς το όσο μπορούμε περισσότερο περαιτέρω πρέπει να είμαστε σε πιο στενή επαφή με την διαμεσολαβήτρια βέβαια και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να την προσκαλέσουμε να έλθει στον, στην Frontex στο άμεσο μέλλον. Το δικό μου μήνυμα όμως που θέλω να σας διαβιβάσω είναι <clears throat> ότι από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η διαδικασία μεταρρύθμισης του κανονισμού της Frontex και η αξιολόγηση για το άρθρο 33 συνεχίζεται. Όλα αυτά σημαίνουν στο μέλλον θα υπάρξει και μια πρόταση τροποποίησης του κανονισμού της Frontex. Θα ήταν καλό για όλους μας αν υπάρξουν συγκεκριμένες και σαφείς ρήτρες που βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, στον κανονισμό αυτό, που θα δεσμεύουν όχι μόνο το φορέα, που αυτό είναι το εύκολο βέβαια, αλλά θα διευκρινίσουν και το ρόλο των ευρωπαϊκών φορέων και συγκεκριμένα της Frontex έναντι των κρατών μελών. Ε, τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να λάβουν υπόψη πολύ σοβαρά τα θέματα της κυριαρχικότητά τους όταν πρόκειται γενικά για την ε, εφαρμογή του νόμου και της τάξης και κυρίως για την προστασία των συνόρων τους μέσα στην συνεργασία με την Frontex. Ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις σας. Και από το Frontex έχουμε και την κυρία Ιγη και τον κύριο Κέσλερ, συμπροέδρους του Συμβουλευτικού Φόρουμ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα για τα θέματα του Frontex. Θα μας παρουσιάσετε τη γνωμοδότηση του Φόρουμ για τα θέματα του Frontex και παρακαλώ περάστε στην παρουσίασή σας Προσπαθήστε να κατανέμετε το χρόνο μεταξύ σας. Όποιος θέλει, ξεκινήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτή την πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Λίμπερ. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το Συμβουλευτικό Φόρουμ μπορεί να σας απευθυνθεί ως Συμβουλευτικό Φόρουμ για θέματα του Frontex. Ο αναθεωρημένος κανονισμός του Frontex προβλέπει αυτήν την ε, μέρημνα για το Συμβουλευτικό Φόρουμ που μπορεί να παράσχει συμβουλές προς το Frontex, τον Frontex, βάσει των όσων τότε επιθυμήσατε και της τότε δέσμευσής σας. Θελήσαμε λοιπόν να δώσουμε συμβουλές στο Frontex ε, για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είμαστε 15 οργανισμοί, σύλλογοι πολιτών, ενώσεις πολιτών και οργανισμοί που ασχολούνται γενικώ με την παρακολούθηση των ανθρωπινών δικαιωμάτων, όπως ο δικός μου. Ε, ακόμη και νομίζω ότι είναι σημαντικό η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και προσφύγων είναι μια κοινή μέρημνα όλων αυτών των οργανισμών που συμμετέχουν στο Συμβουλευτικό Φόρουμ του Frontex. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την πρόσβαση σε πραγματικά ένδικα μέσα και εδώ καλωσορίζουμε την στήριξη της έκκλησης της ευρωπαϊκής Δημοσιολαβήτριας να κοιτάξουμε καλύτερα το πώς αυτό μπορεί όντως να λειτουργήσει στην πράξη και στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του Frontex. Ο, η διαμεσολαβήτρια έχει σωστά επισημάνει ότι ο Frontex παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την σωστή πρόβλεψη προτύπων με όλες του τις επιχειρήσεις. Συμφωνούμε για τη διάκριση μεταξύ των δράσεων εντοπισμού και των προσφυγών, των διαδικασιών προσφυγών. Δεν μπορεί το ένα να αντικαταστήσει το άλλο, πρέπει και τα δύο να αντιμετωπιστούν με τη δέουσα προσοχή. Η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης είναι από τις βασικές λειτουργίες του Frontex, διότι ο υπεύθυνο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Frontex κοιτάζει να δημιουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό και βρίσκεται σε στενή επαφή και ε, συνομιλίες με το Συμβουλευτικό Φόρουμ. Στην ουσία, μιλούμε για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο αποτελεσματικό και ε, χειροπιαστό σύστημα μετά από ένα χρόνο εμπειρίας. Επίσης, όπως σωστά σήμερα ο διευθυντής του Frontex, τι μπορεί να κάνει ο Frontex για να φέρει πέρα στις ευθύνες του, να παράσχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να δημιουργήσει ένα μηχανισμό που επιτρέπει την ε, πρόθεση των ε, προσφυγών των μεμονωμένων προσώπων. Μιλάμε για παραβιάσεις θεμελιδών δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις κοινέ επιχειρήσεις του Frontex για τέτοιου είδους υποθέσεις. Δεν θα παρουσιάσω τις διάφορες υποθετικές καταστάσεις όταν μιλάμε για κοινέ επιχειρήσεις του Frontex. Ο κοινωνιστικός διευθυντής σωστά σας επεσήμανε κάποιες από τις περιπτώσεις, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες υποθετικές καταστάσεις που σας ανέφερε είναι σωστές. Μιλάμε για το προσωπικό του Frontex, για διερμηνείς, για αξιωματικούς, για αποσπασμένους, εργαζομένους και το καθεξής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν μιλάμε για περιστατικά ή για προσφυγές που αφορούν προσωπικό ή αξιωματικό του Frontex, τότε είναι ευθύνη του Frontex να ασχοληθεί με την προσφυγή. Αυτό είναι αναντήρητο. Όμω, εάν τα κοιτάξετε προσεκτικότερα και δείτε όλε τι υποθετικέ καταστάσει που σα ανέφερε και ο εκτελεστικό διευθυντή, θα καταλάβετε ότι είναι προφανέ οι προσφυγέ των μονομένων ατόμων κατά προσώπων που δεν ανήκουν στο προσωπικό του Frontex μπορούν τελικά μόνο εφόσον υπάρξει προσφυγή σε επίπεδο κρατών μελών, στις αρχές των κρατών μελών να εξεταστούν. Είναι λοιπόν καθοριστική σημασία όταν δημιουργεί το μηχανισμό παρακολούθησης ο Frontex να λαμβάνει υπόψη και το κατά πόσο μπορούν να αναλάβουν εδώ ρόλο και τα κράτη-μέλη στην εξέταση των ατομικών προσφυγών, ώστε να υπάρξουν ανεξάρτητες και ε, πραγματικές έρευνες, ανακρίσεις. Αυτό είναι σημαντικό για το μηχανισμό παρακολούθησης, διότι μόνο έτσι μπορεί να καθοριστεί ε, ο ρόλος των μεν και των δε και να υπάρξει και η ανάλογη διαδικασία. Συνοπτικά, πρόκειται βεβαίω για ένα θέμα αρκετά περίπλοκο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο εδώ, αλλά ο συνάδελφο ο κ. Κέσλερ θα συνεχίσει νομίζω λίγο από αυτού. Νομίζω ότι ως συμπρόεδρος του Συμβουλευτικού Φόρουμ θα ήταν καλό να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία του παρουσία τη Ευρωπαϊκή Διαμεσολαβήτρια, για να ακούσει και ο εκτελεστικό διευθυντή. ότι κάποιε προσφυγέ πρέπει να γίνονται και υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια στηρίζει αυτή την εκδοχή. Αλλά εδώ μιλάμε για ατομικέ προσφυγέ όπου ο προσφεύγων δεν είναι ούτε το θύμα, ούτε του έχει δοθεί η εντολή να προσφύγει από κάποιο θύμα. Το θέμα είναι απλώ το κατά πόσο υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για ένα περιστατικό. Αυτό πρέπει να καταστεί σαφέ για να γίνει σωστή διάκριση από τι γενικές προσφυγές κατά της μεταναστευτική πολιτικής της Ευρωπαίας Ένωσης και ε, των ε, κανόνων που προκύπτουν για τα θεμελιώδη δικαιώματα με τι ατομικέ προσφυγέ. Για το μηχανισμό το, της εξέτασης των προσφυγών. Ο Frontex θα μπορούσε να συνεχίσει να ενθαρρύνει και επιμένω αυτό, θα μπορούσε να συνεχίσει να ενθαρρύνει την καταγραφή περιστατικών και τις προσφυγές σε κοινέ επιχειρήσεις. Ο Frontex θα μπορούσε να παράσχει πληροφορίες για τις προσφυγές που αφορούν το προσωπικό του Frontex, τους απεσταλμένους αξιωματικούς, και σε γλώσσα που να είναι κατανοητή για τους μετανάστες επίσης. Θα θέλαμε ο Frontex να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές της ανακρίσης και την εξέταση των προσφυγών. Ακόμη, ο Frontex θα μπορούσε να συνεργάζεται με τους εθνικούς διαμεσολαβητές και τους εθνικούς φορείς που ασχολούνται με τα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής για να γίνεται σωστή εξετάση των προσφυγών θα πρέπει ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής να ασχολείται με τις προσφυγές που γίνονται για το προσωπικό του Frontex και διεθνώς να υπάρχει εξετάση των προσφυγών αυτών από τους υπόλοιπους διαμεσολαβητές. Ο διευθυντής του Frontex θα μπορούσε εκ μέρους του οργανισμού να λαμβάνει και να εξετάζει αυτές τις προσφυγές αξιοποιώντας όλους τους ανθρωπίνους πέρος πόρους που υπάρχουν. Με τις υπάρχουσες προβλέψεις δεν θα μπορέσει να φέρει πέρα σε αυτή την αρμοδιότητα. Το θέμα είναι πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια που υπάρχουν. Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης στην Μεσόγειο, για την ώρα δεν είχαμε προσφυγές από μετανάστες ε, σε περίπτωση εθνικών επιχειρήσεων όπου δεν ήταν παρόν ε, ο Frontex αλλά θα πρέπει και αυτού του είδους οι προσφυγές να μπορούν να εξεταστούν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κέσλερ. Είστε μάρτυρας ότι για πρώτη φορά ε, ακούσαμε το Συμβουλευτικό Φόρουμ. Είναι η πρώτη φορά που ήρθατε. Και εσεί το ίδιο, κύριε Γιουγκέγκορ, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε το ίδιο το συμβουλευτικό φόρουμ. Ακούμε εσά μόνον πρώτη φορά. Ακούσαμε λοιπόν τις παρουσιάσεις του της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, του Διευθυντή του Frontex και του Συμβουλευτικού Φόρουμ. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θα θέλετε το λόγο. Θέλετε να κάνετε σχόλια. Κάποιος, κανείς. Θα ήθελα να δω χέρια να υψώνονται. Ωραία. Βλέπουμε ότι υπάρχει συμμετοχή. Κύριε Μπρόγκς, μπορείτε να ξεκινήσετε. Είστε ο πρώτο που είπε το λόγο. It's customary. Ευχαριστώ. Ήθιστε να λέμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα και θα πρέπει να γίνονται σεβαστά όλα από όλους. Κάποια από αυτά είναι προφανές ότι ισχύει αυτό. Για παράδειγμα, ότι μιλάμε για την απαγόρευση των βασανιστήριων ή τη σκληρή απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση. Προφανώ. Ωστόσο, ίσως κάποια πρόσωπα εξαιτία τη συμπεριστοφοράς του ή τη υπόνοια για συγκεκριμένη συμπεριφορά που έχουμε μπορεί να θέσουν τον εαυτό του σε μια κατηγορία στην οποία επιφυλάσσουμε διαφορετική μεταχείριση. Για παράδειγμα, όταν κάποιο από μόνο του τοποθετεί τον εαυτό του στην κατηγορία των ε, παράνομων μεταναστών, παράτυπων μεταναστών, αμέσω χάνει το δικαίωμα τη ελεύθερη μετακίνηση εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αξιωματούχοι λοιπόν της Frontex και των κρατών μελών θα πρέπει να ασκούν ε, καταναγκαστικά μέτρα όταν διεξάγουν μία ανάκριση αυτών των προσώπων, όταν για παράδειγμα υπάρχει πλαστογραφία ή καταστροφή εγγράφων πρέπει να υπάρχει και κράτηση και να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Αναφέρθηκε η διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα και προφανώς και εγώ υποστηρίζω ότι έχουμε καθήκον να σώζουμε κάποιον στην θάλασσα. Ωστόσο είναι διαφορετικό το να τους σώσουμε από πνιγμό και χωρίς να τους ανταμείψουμε με το να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μπουν στην Ευρώπη πρέπει να τους στείλουμε πίσω στη χώρα τους. Γιατί συχνά τους δίνεται δυνατότητα παραμονής. Έχουμε ένα περιστατικό νομίζω πριν δύο χρόνια ότι όταν δεν τους δίνεται άσυλο, τους δίνεται απλώς ένα, μια διαταγή απέλασης στην οποία ευγενικά τους ζητούμε να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να αναγκαστούν να ε, επιστρέψουν στη χώρα καταγωγή τους. Δεν θα ήθελα η Frontex να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των ε, κακόβουλων καταγγελιών. Θα, προσωπικά θα πίστευα ότι θα ήταν σκόπιμο να καταγράφουμε με βίντεο ε, πάντα τις όποιες ε, επαφές του μεταξύ των ε, αξιωματικών που, και των αστυνομικών και των μεταναστών. Γιατί Συχνά οι καταγγελίε, αν κατάλαβα καλά, δεν γίνονται από τους ίδιους τους μετανάστες, αλλά από μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο όνομά τους, χωρίς να τους έχουν προ τούτο εξουσιοδοτήσει οι μετανάστες. Στο αστικό δίκαιο, οι εργοδότες ευθύνονται για την ε, πράξεις και τις παραλήψεις των εργαζομένων τους, γιατί έχουν τη δυνατότητα να τους απολύσουν. Ωστόσο δεν ευθύνονται για πράξεις ανθρώπων επί των οποίων δεν ασκούν κανέναν έλεγχο. Επομένως, μου φαίνεται απαράδεκτο, ε, αδιανόητο η Frontex να έχει ε, ευθύνη για τις ε, δράσεις των ατόμων που, των κρατών μελών. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ. Αισθάνομαι κάπως μοναχικά έχοντας ακούσει τις τέσσερις παρουσιάσεις. Γιατί, ποιο είναι το θέμα εδώ. Φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν παραχωρήσει ε, μια δραστηριότητα που ήταν δικιά τους αρμοδιότητα αρχικά, δηλαδή την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή, ε, ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που αναλαμβάνει αυτή την αρμοδιότητα μας λέει ότι δεν μπορεί να αναλαμβάνει την ευθύνη όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά, ε, παραπέμπει στα κράτη-μέλη και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μας λέει ότι αυτό δεν είναι δυνατό. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε επιτόπου ε, αστυνομικούς που να φέρουν στολή με την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερθήκατε και στη σχετική νομολογία του δικαστηρίου, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτοί οι αξιωματικοί δεν φέρουν καμία ευθύνη, είναι εκτός ε, δημοκρατικής λογοδοσίας. Επομένως έχουμε κάνει πλέον παραχώρηση όχι μόνο της αρμοδιότητας της επιτήρησης, έχουμε παραχωρήσει και τις ευθύνε. Καταλαβαίνω ότι ο διευθυντής μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας από μόνος του δεν μπορεί να το λύσει, αλλά πριν λίγο μόλις είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων για το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου για την διάσωση στη θάλασσα, για την εντολή της Frontex, τι μπορεί να γίνεται και τι μπορεί να γίνει. Και λοιπόν το ερώτημα που θέτω σε όλους είναι, ωραία, και μετά από όλα αυτά τι, τι περιθώριο ελιγμών έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι τελικά θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα είναι αρμόδιος, θα έχει την ευθύνη να φροντίζει τη μεταχείριση των προσφύγων και, στον, και από τον οποίο θα ζητηθεί λογοδοσία όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Επίσης, το ζήτημα που έθεσε ο κύριος ε, Κέσλερ για το ποιος μπορεί να κάνει μια καταγγελία, ποιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μια καταγγελία. προφανώς, εάν έχει κάποιο διαφορετική άποψη για τον κανονισμό του Βλήνο 2 ή για το, την επαναπρόθεση ή οποιαδήποτε ε, νομοθεσία ευρωπαϊκή, δεν θα υποβάλει καταγγελία στη Frontex, αλλά εάν ένας μετανάστης ή αν μία μη κυβερνητική οργάνωση σκοπεύει να κάνει ομαδική προσφυγή, θα πρέπει να γνωρίζει προς ποιον μπορεί, και εναντίον ποιου μάλλον μπορεί να προσφύγει. Και αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύρια Οράιλη, είπατε ότι θέλετε να υπάρχει ένας εσωτερικός μηχανισμός υποβολής παραπώνων στην Frontex. Και στο τέλος της παρουσιάσεως σας αναφερθήκατε στην ε, τραγωδία της Λαμπεντούζα που χάσανε τη ζωή τους εκατοντάδες άτομα. Αυτό όμως μας οδηγεί σε πολλά ερωτήματα, τουλάχιστον σε μένα. Κάπου υπάρχει η ιδέα σε ορισμένους, στη σκέψη ορισμένων ότι η Frontex ήταν υπεύθυνη για τους ε, θανάτους αυτούς των εκατοντάδων ατόμων. Αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο πιστεύω να το πιστεύει κανείς. Αν υποβληθούν παράπονα, τι θα κάνετε με αυτά τα παράπονα. Εγώ πήγα στην Ισπανία για να δω πώς λειτουργεί εκεί η Frontex. Είδα την καθημερινή τους λειτουργία πώς λειτουργεί σε καθημερινό επίπεδο η Frontex και μιλήσαμε με πολλά άτομα εκεί. Μιλήσαμε με αυτούς που είχαν έρθει από τη Βόρεια Αφρική και είχαν περάσει τα στενά του Γιβραλτάρ, με αστυνομικούς, με μέλη της Frontex. Αυτό το οποίο προήλθε από όλες αυτές τις συζητήσεις ήταν ότι πολλά άτομα τα οποία δεν έχουν τα προαπαιτούμενα για να πάρουν το καθεστώς του πρόσφυγα, ψεύδονται για να μπορέσουν να διεκδικήσουν έτσι κι αλλιώς ένα καθεστώς ασύλου, ένα καθεστώ πρόσφυγα σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λάβουμε λοιπόν αυτό υπόψη, με ποιο τρόπο θα προστατεύσετε το προσωπικό της Frontex από ψευδείς καταγγελίες που γίνονται εναντίον τους. Θέλετε να έχετε ένα εσωτερικό μηχανισμό υποβολής παραπώνων. Πώς θα αποφύγετε όμως, πώς θα αποτρέψετε την κατάχρηση αυτού του συστήματος από άτομα τα οποία ζητούν το καθεστώ του πρόσφυγα, γιατί το κάνουν προφανώς για να μπορέσουν να μείνουν στο έδαφο του κράτου μέλου, όπου γίνεται αυτό. Όπως είπε και η κυρία Σατζεντίνη, και εγώ πρέπει να εκφράσω την ευρωοντιστία μου ενώπιον τη κατάστασης όπως έχει παρουσιαστεί σήμερα. Και δεύτερον θέλω να πω ότι έχω την εντύπωση ότι ο ενθουσιασμός μας είναι λιγάκι πιο περιορισμένος σε σχέση με την προηγούμενη ακρόασή μας σε ό,τι αφορά την βελτίωση που έχει επέλθει μετά την τροποποίηση του κανονισμού της Frontex. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι κατανοώ αυτή τη στιγμή είναι ότι το θέμα αυτό για την υποβολή παραπώνων είχε αναφερθεί προηγουμένως στη διαδικασία μεταρρύθμισης. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί αρκετά σε βάθος για να μπορούμε να έχουμε τι κατάλληλε κατευθυντήρες γραμμέ, οι οποίε είναι στενάρε και να μπορέσουμε να διαλύσουμε τι παρεξηγήσει και τι αμφισημίε σε αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω τώρα αν εμεί πέντε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορέσουμε να δώσουμε μια οριστική λύση για τα θέματα αυτά. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να υπάρξει και κάποια συζήτηση και πρόοδος για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί και για να μπορέσουμε να βγούμε από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω συγκεκριμένα ιδέες. Και τώρα επανέρχομαι στους ομιλητές μας. Ακούσαμε τις απόψεις των ε, βουλευτών για το θέμα αυτό και ακούσαμε φυσικά και αυτά που είπε ο Διευθυντής του Φόρεα και η διαμεσολαβήτρια. Ίσως θέλετε να κάνετε περαιτέρω σχόλια ή απαντήσεις σε αυτά που ακούσατε από τους βουλευτές. Έχετε το λόγο σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία τον λογο σας ευχαριστω πολυ λεει η κυρια οραιλη Ευχαριστώ για τα ερωτήματα και τις ε, παρατήρησεις σας. Τα έχω καταγράψει όλα αυτά, διότι καταδεικνύουν πόσο απαραίτητο είναι να δημιουργηθεί ένας εσωτερικός μηχανισμός επεξεργασίας παραπώνων. Έχουμε ακούσει για την πολυπλοκότητα του συστήματος, ακούσαμε για την επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ κατών μελών Frontex και άλλων φορέων. Για μένα όμως η δημιουργία ενός σωστά λειτουργούντο λειτουργούντος ανεξάρτητου και με εμπειρογνωμοσύνη μηχανισμού παραπώνων θα μας επέτρεπε να διαλύσουμε αυτό το νεφέλωμα μέσα στο οποίο κινούμαστε σε ό,τι αφορά και τις επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει τώρα ένα καταπληκτικό μηχανισμό αντιμετώπισης παραπώνων, σαν παράδειγμα, και αντιμετώπισε τις ίδιες δυσκολίες που αναφέρθηκαν εδώ σε σχέση με τις ε, δραστηριότητες της εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόρεσε να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και να ξεπεράσει όλες αυτές τις αρχικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή και θέλω να προσκαλέσω τον κύριο Λάιτινεν και την Frontex να συνεργαστούν μαζί μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια από αυτά τα προβλήματα και να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το οποίο επέτυχε να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις κακόβουλες καταγγελίες όπως είπε ο κύριος Κλάις. Αυτό είναι κάτι που έχει να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε φορέα που δέχεται παράπονα ή οποιοδήποτε διαμεσολαβητή. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διαμεσολαβητέ αστυνομίας που αντιμετωπίζουν παράπονα που υποβάλλονται για τι αστυνομικέ αρχέ των κρατών μελών και έχουν την εμπειρογνωμοσύνη, θα έπρεπε να έχουν την εμπειρογνωμοσύνη και τους θεσμικούς πόρους και τη θεσμική πείρα και ευφύεια για να μπορούν να διακριβώσουν ποια παράπονα είναι κακόβουλα και ποια είναι εδρεωμένα. Και αυτό είναι μια δυνατότητα σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης. Αν έχετε όμως ένα μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί, αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κατανοώ αυτό που λέει και ο κύριος Μπρόνς <clears throat> σε σχέση με την έλευση εγκληματιών που έρχονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι οποίοι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο ευγενείς και αυρόφρονες ώστε να εξηγούν για ποιο λόγο έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι όμως νομίζω ότι το να υπάρχει ένα σωστά λειτουργούν, λειτουργών μηχανισμός παραπώνων με την απαραίτητη χρηματοδότηση θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα θέματα αυτά. Επίσης ό,τι αφορά την αρμοδιότητα και την ευθύνη των κρατών μελών. Ένα από τα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει έτσι η Frontex είναι ότι αν διαπιστώσει κάποια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πλευρά των κρατών μελών κατά τη διάρκεια μιας κοινή δράσης είτε είναι ε, επαναπροώθηση ή απόθεση οτιδήποτε, να έχει τη δυνατότητα η Frontex να κάνει ένα παράπονο προς την Κομισιόν σε σχέση με μια παραβίαση των συνδικών και η Κομισιόν θα έπρεπε να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Δηλαδή ο μηχανισμός εσωτερικής υποβολής παραπώνων είναι ένας τρόπος να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό σας προτείνω να εργαστούμε από κοινού και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά όλοι μαζί. Τελικά θα βοηθήσει πάρα πολύ το θεσμό της Frontex. Ευχαριστούμε κύριε Λάιτινεν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής σας για τα σχόλιά τους. Είναι πολλά τα ζητήματα που επανέρχονται κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Ε, ας δούμε πρώτα το τι έχει έρθει στα χέρια μας ως ε, παράπονο, ω προσφυγή ως τώρα. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των ε, προσφύγων που έχουμε λάβει αφορούν τις συνθήκες κράτησης ε, στα κάτι μέλη. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις ε, επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα. Ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν εδώ. Μιλήσαμε, μιλήσατε και με τον αφορμή του, την έκθεση του κυρίου Κοέλιου για τους κανόνες που πρέπει να διέπουν αυτές τις περιπτώσεις διάσωσης. Τρίτη ομάδα, όχι μικρότερη, είναι οι επικριτικές, τα επικριτικά σχόλια για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για τις επιστροφές, είτε για την μετανάστευση γενικότερα. Και εμείς είμαστε στην εχνή αυτών των επικριτικών σχολείων. Υπάρχουν και μεμονωμένες όμως περιπτώσεις και αυτό νομίζω είναι ακριβώς το σκέλος το οποίο συζητάμε. Έχουν υπάρξει οι απόπειρες να εξαντληθεί το δυναμικό του οργανισμού σε ορισμένες κατηγορίες προσφυγών. Σωστά αναφέρατε εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν φτάνουν στα χέρια μας τέτοιες προσφυγές, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όσο το περισσότερες πληροφορίες γίνεται από τα ενδιαφερόμενα, από τα οικία κάτι μέλη, με διαφορετικό βαθμό επιτυχίας. Κάποιοι είναι πιο λεπτομερείς στις απαντήσεις τους, κάποιοι δρούν ε, πολύ γρήγορα, έγκαιρα, κάποιοι όχι, αλλά εκεί πρέπει να υποβληθούν όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Δεν ανέφερα ειδικό στον κώδικα συμπεριφορά για τις κοινέ ε, επιχειρήσεις επιστροφής. Όμως, όταν αναφέρθηκαν οι επιστροφές, είναι και αυτό ένα άλλο εργαλείο, ένα άλλο μέσο που αναπτύξαμε σε καλή συνεργασία με το Συμβουλευτικό Φόρουμ. Αυτό εν μέρη αντικατοπτρίζει και τις ανάγκες που καλούμαστε να καλύψουμε. Έχουμε εξετάσει κατά το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τις προσφυγές. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Είναι ένα ενδιαφέρον σύστημα και πραγματικά κοιτάζουμε πώς θα μπορούσε να, μας, ε, να προσαρμοστεί και στις δικές μας ανάγκες. Αντί όμως το να μένουμε στα προβλήματα που είχαμε ως τώρα και τις προκλήσεις μόνον και παρακαλώ μην με παραρμηνεύσετε, θα ήθελα να κοιτάζουμε και πέραν των μηχανισμών για τις προσφυγές, για τα παράπονα, διότι αυτό που διαρκώς απαντούμε ξανά και ξανά ως εμπόδιο είναι ο ρόλος των κρατών και η προθυμία τους να δώσουν πρόσβαση στον Frontex σε κάποιες πληροφορίες. Αυτό το σημείο μπορεί να επιληθεί μόνο αν υπάρξουν σαφείς διατάξεις. Με άλλα λόγια, εάν δημιουργηθεί νόμος. Νόμος ο οποίος υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στον χειρισμό αυτών των θεμάτων μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να κοιτάξουμε λίγο παραπέρα, όχι μόνο τον μηχανισμό των προσφύγων αυτών καθεαυτών, διότι μπορεί να δώσει διαφορετικού είδους αποτελέσματα ούτως ή άλλως, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο ρόλος των κρατών μελών. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και θα ήθελα η επόμενη τροπολογία του κανονισμού του Frontex να το συμπεριλάβει. Νομίζω δηλαδή πιο σωστό είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να έχουμε κάποιες επιπλέον εξελίξεις να επιλύσουμε κάποια ζητήματα παρά να αναφέρουμε μόνο προβλήματα και να λέμε το ένα και το άλλο είναι ανέφικτο. Δεν είναι ανέφικτο. Έχουμε δεσμευτεί να εξεύρουμε λύσεις. Αλλά πρέπει να καταλάβετε όλη την εμβέλεια του προβλήματος και το διαφορετικό ρόλο που παίζουν όλοι οι συμμετέχοντες σε τέτοιες καταστάσει. Ευχαριστούμε από το Συμβουλευτικό Φόρουμ. Θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Απλώς να θυμίσω και πάλι τώρα που βλέπουμε καλύτερα πώς εργάζεται ο Frontex, επειδή συνεργαζόμαστε εδώ και 1,5 χρόνο, νομίζω είναι σημαντικό να μην βλέπουμε μεμονωμένα τις επιχειρήσεις του Frontex. Διότι αυτό που εγώ και ο Στέφαν αναφέραμε ήδη είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό ακριβώς να δούμε τις υπάρχουσες δομές των κρατών μελών, διότι έχουν τα δικά τους ιδρύματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικά τους, τους δικούς τους φορείς διαμεσολαβητών, αυτά υπάρχουν. Και ο παραδοσιακός τρόπος που προωθεί ο Frontex τις ατομικές προσφυγές σε συνεργασία μόνο με τις εθνικές αρχές ίσως να μην είναι η καλύτερη λύση για το μέλλον. Αυτό είναι μια πρόσθετη ιδέα από δικής μας πλευράς. Μια νέα ιδέα που ε, υπονοεί ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις υπάρχουσες εθνικές δομές και να είναι πιο αποτελεσματικές στις ανακρίσεις και την επιβολή κυρώσεων και την αποζημίωση κάποιων θυμάτων. Κύριε Κέσλερ, Μια σύντομη απάντηση σε μια από τις ερωτήσεις ενός βουλευτή. Δεν μιλάμε για δικαστικές προσφυγές που υποβάλλονται στο Frontex ως δικαστικό φορέα, ως δικαστικό σώμα. Κάθε δημόσιος φορέας που χρεούται να διεξαγάγει ανάκριση σε περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αδίποτε πληροφορία προέρχεται από παρατηρητή ο οποίος δεν έχει λάβει σχετική διαταγή όπως από μια μη κυβερνητική οργάνωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και από τον ίδιο το Frontex ή από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Αυτό εννοούσαμε και να σας θυμίσω ότι το καθεστώς του μετανάστη δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει ανθρώπινα δικαιώματα και εδώ μιλάμε για παραβιώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ίσως ένα τελευταίο σχόλιο Ετοιμάζουμε τώρα την ετήσια έκθεση του Συμβουλευτικού Φόρουμ και όπως είπε η Άινταν, έχουμε ένα χρόνο περίπου που λειτουργούμε. Η έκθεση αυτή λοιπόν θα παρουσιάζει το έργο μας ω τώρα και ευχαριστώ να σας, την παρουσιάσουμε μόλι είναι έτοιμη και πρόκειται να δημοσιευτεί. Thank you. Thank you. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για τι ε, παρουσιάσεις και τα σχόλιά σα. Άλλες παρεμβάσεις από του συναδέλφου, όχι, ωραία. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ράιλι για την παρουσίασή τη τον κύριο Λάιτινεν τους εκπροσώπους του Συμβουλευτικού Φόρουμ θα έλεγα σε λίγα λεπτά και να περάσουμε και στο επόμενο σημείο. Δύο λεπτά νωρίτερα. Ξαναρχίζουμε. Συνεχίζουμε με το σημείο που ήταν προγραμματισμένο στις 11. Ε, Συνεχίζουμε με αυτό το σημείο, λοιπόν, γιατί είναι σχεδόν 11 παρουσίαση τη μελέτη υπό τη διαχείριση τη μονάδα εκ των προτέρων εκτίμηση αντικτύπου σε συνεργασία με το τμήμα πολιτική για την εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης των προσώπων. Θα ακούσουμε την ε, Μιλιέ LTD. Μονάδα εκ των προτέρων εκτίμησης αντικτύπου σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Γάμα, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Θα θυμάστε ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ το 2012 ζήτησε να εκπονηθεί μελέτη αντικτύπου για την προτινόμενη οδηγία για την ίση μεταχείριση η μελέτη συντάχθηκε από, το, από τη συμβουλευτική μιλιά και την εξέτασε η μονάδα σε συνεργασία με το τμήμα πολιτικής που προανέφερα. Έχει μοιραστεί. Η αρχή, η μελέτη, μελετή, μελετά την υλοποίηση της αρχής τη ίση μεταχείριση των προσώπων, ασχέτω ε, προέλευση, καταγωγή, ε, σεξουαλικών προτιμήσεων, υγεία ή αναπηριών. Σήμερα θα έχουμε την παρουσίαση τη μελέτη και απλώ να εκφράσουμε την ε, δυσαρέσκειά μα που εδώ και χρόνια, τέσσερα χρόνια, ξεκινήσαμε να συζητάμε το θέμα αυτό και παρέμενε εκκρεμέ. Επί χρόνια η οδηγία τη ίση μεταχείριση είναι μπλοκαρισμένη στο Συμβούλιο. Θυμάμαι πολύ καλά όταν ξεκινήσαμε το 2009 ήταν μία από τις πρώτες προτεραιότητες της ε, νέο εκλεγήσεως ε, επιτροπής. Κάποιοι από εμάς τότε είχαμε επιμείνει με τα υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε απευθυνθεί μέχρι και στον πρόεδρο Μπαρόζο ε, για να προχωρήσει η οδηγία αυτή, για το καλό όλων. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Η οδηγία για την ίση μεταχείριση παραμένει μπλοκαρισμένη στο Συμβούλιο επί σειρά τεσσάρων ετών. Αυτό πραγματικά είναι κρίμα. Οπότε έτσι ενισχύεται η πεποίθησή μας ότι είναι πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται σε κρίση, όχι μόνο το ευρώ και η οικονομική διαχείριση, αλλά και η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αξίες και αρχές, σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ισότητα έναντι του νόμου ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Λέβεντ Άλτεν, ο οποίος είναι επιστημονικός συντονιστής για την μελέτη για τι μελέτε αντικτύπου και μετά θα ακούσουμε τους σχεώδεις μας τους εισηγητές και σκιώδεις μας για τα σημεία που μας ενδιαφέρουν. Θα δώσουμε βεβαίως το λόγο και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Προεδρίας. Πρώτα, ο λόγος στην μονάδα για τις μελέτες αντικτύπου. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους. Έχω μια παρουσίαση περίπου 10 λεπτών. Θα είμαι σύντομος. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν το πεδίο εφαρμογή και τους στόχους που θέσαμε στην μελέτη, δηλαδή ποιες περιοχές εξετάσαμε, δεν τα εξετάσαμε όλα. Και μετά, λίγο πιο λεπτομερικά, τα αποτελέσματα της μελέτης και κάποια συμπεράσματα. Πρώτον, όσον αφορά το πεδίο της μελέτης. Τι εξετάσαμε. Δεν εξετάσαμε τα πάντα. Αυτά που μας ζητήθηκε ήταν να εξετάσουμε το κόστος και το όφελος και για τις δημόσιες αρχές, καθώς επίσης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή δεν εξετάσαμε το ζήτημα. Μάλλον εξετάσαμε το ζήτημα για την κοινωνία συνολικά και αυτός ήταν ο στόχος της έκθεσης. Αυτό το πεδίο μελέτης προέκυψε αφενός ε, εξαιτία των ανησυχιών που έχει εκφράσει το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, οδηγία, καθώ επίση και η ανησυχία που έχει εκφραστεί για το γεγονό ότι δεν έχει αξιολογηθεί το αποτέλεσμα και οι επιπτώσει τη ε, νομοθεσία που ήδη υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω σε σχέση με το ζήτημα τη επικούρικότητα των συστημάτων πρόνοια. Υπάρχουν επίση ανησυχίε όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου, ιδίως σε σχέση με συγκεκριμένα άρθρα αλλά επίσης και το κόστος που επιβαρύνει το δημόσιο προπολογισμό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, η Επιτροπή έχει ήδη αξιολογήσει εκτενώς, έχει ήδη εξάγει μια εκτενή αξιολόγηση αντικτύπου την οποία αξιοποιήσαμε. Είχαμε πολλά στοιχεία από εκεί. Εκεί εξετάζεται λεπτομεριακά το ζήτημα του ποιο είναι το όφελος και ποιο είναι το κόστος για την κοινωνία συνολικά. Εμείς περιληπτικά αναφερόμαστε στο θέμα, δεν πηγαίνουμε λοιπόν σε μεγαλύτερο βάθος στο ζήτημα της κοινωνίας συνολικά. Εμείς εστιαστήκαμε στους δύο τομείς που προείπα. Εάν κανείς εξετάσει συνολικά το θέμα, θα, έλεγε, θα λέγαμε ότι η έκθεση δική μας συμπληρώνει την έκθεση της Επιτροπής και την αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής. Όσον αφορά την προσέγγιση που ακολουθήσαμε, τη μεθοδολογία, όπως είπα δεν μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τα πάντα. Η οδηγία καλύπτει πάρα πολλού τομεί και πολλές μορφές διακρίσεων. Επομένω, επιλέξαμε εκείνες τις περιοχές τις οποίες αν αναλάβουμε δράση θα έχουμε το μεγαλύτερο όφελος ή θα είναι εφικτό να μειώσουμε κατά το μεγαλύτερο βαθμό το κόστος δηλαδή τις περιοχές εκείνες που είναι πιο σημαντικές. Και δεν ε, ασχοληθήκαμε με περιοχές που ε, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας, όπως για παράδειγμα η ε, ειδική αγωγή, η παροχή υπηρεσιών πρόνοιας σε συγκεκριμένες ομάδες. Επίσης, εστιάσαμε στους τομείς εκείνους όπου οι διακρίσεις είναι πιο έντονες η, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας, εξάλλου η οδηγία ζητά να εστιάσει το δράση του, κράτους μέλος στους τομείς εκείνους όπου μπορεί να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να αξιολογήσουμε, να εκτιμήσουμε πόσο θα είναι το, το κόστος και το όφελος μιας συγκεκριμένη δράση σε ένα κράτος μέλος. Είδαμε τι έχουν κάνει άλλα κράτη-μέλη, αλλά Αξιοποιήσαμε επίσης και τη διεθνή εμπειρία. Και, ε, κυρίως κράτη τα οποία έχουν βέλτιστες πρακτικές όπως η Αυστραλία ή οι Ηνωμένε Πολιτείε που έχουν χρόνια εμπειρίας στην υιοθέτηση και την εφαρμογή νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων ιδίω κατά των ατόμων με αναπηρία. Επίσης θέλαμε να βασιστούμε σε υφιστάμενα δεδομένα ε, όλες αυτές οι παράμετροι μας οδήγησαν στην επιλογή των ε, τομέων που τελικά αξιολογήσαμε. Οι τομεί αυτοί λοιπόν είναι το κόστος, το διοικητικό κόστος και το κόστος των διαχειριστικών αρχών, των ελεγκτικών αρχών, δηλαδή κόστη τα οποία ε, επομίζεται το κράτος που δημιουργεί τέτοιους ε, μηχανισμούς ε, είτε που ελέγχουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, είτε που ευαισθητοποιούν το κοινό. Το κόστος των υπηρεσιών παροχής, των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας ή επίσης ε, ε, εξετάζουν καταγγελίες ή νομικές προσφυγές και μετά δράσεις που μπορούν να αναλυφθούν σε συγκεκριμένους τομείς, δηλαδή για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσει σε συγκεκριμένους τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία κτλ. Και όσον αφορά το όφελος, εμείς όπως σας είπα εστιάσαμε στο όφελος που θα είχαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι γενικά η κοινωνία. Η... Τα ίδια τα άτομα με αναπηρία για παράδειγμα, γιατί αυτό ήταν κάτι που κάλυψε η Επιτροπή. για λόγους πρακτικούς ε, ασχοληθήκαμε με πέντε κράτη-μέλη, την Τσεχία, την ε, Γερμανία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Εξετάσαμε λοιπόν ε, ενδελεχώς την κατάσταση σε αυτά τα πέντε κράτη-μέλη. Πράγμα που σημαίνει ότι τα στοιχεία και τα αριθμητικά στοιχεία που θα σας παρουσιάσω αφορούν τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη τις ιδιαιτερότητες αυτών των κρατών μελών τις λάβαμε υπόψη μας. Για παράδειγμα, αν, υπάρχου, αν, αν συχνά στο ραδιοτηλεοπτικό τομέα χρησιμοποιούνται υπότιτλοι για τους κοφούς. Αυτό το λάβαμε υπόψη μας. Ο τομέας ε, στον οποίο χρειάζονται δράσεις οι οποίες θα έχουν σημαντικό κόστος είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων κατά ατόμων με αναπηρία. Ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση, τη στέγαση, τις υπηρεσίες πρόνοιας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή γενικά την πρόσβαση αυτών των ατόμων σε ξενοδοχεία, σε, δημόσια κτίρια κτλ. Το, το, το σημαντικότερο θέμα για τα άτομα με αναπηρία είναι η πρόσβαση σε, κτίρια. Σύμφωνα με το Σύμφωνα του ΙΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, απαιτείται από τα κράτη-μέλη να ε, διευκολύνουν τα άτομα στην ε, συμμετοχή τους στην κοινωνία. Αυτή λοιπόν, λοιπόν ήταν οι κύριοι τομεί που εξετάσαμε σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία. Όσον αφορά τι διακρίσει βάσει την ηλικία, είχαμε δύο ζητήματα που, που εξετάσαμε, του ε, νευροπαθεί και εκείνου που πάσχουν από κατάθλιψη. Καθώ επίση και την ε, Στη, στην περίπτωση των διακρίσεων ε, εξαιτία σεξουαλικού προσανατολισμού εξετάσαμε το ζήτημα της φορολογίας και της, της μεταχείρισης ε, στα περιουσιακά θέματα. Δεν εξετάσαμε ζητήματα που έχουν σχέση με θρησκευτικέ διακρίσεις. Έχετε χρόνο, έχετε χρόνο, καθίσχαζε ο Πρόεδρος. Ωραία, θα, θα, σας δώσω τα αποτελέσματα για καθέναν από τους τομείς που ανέφερα. Για να εξηγήσω και πάλι γιατί δεν εξετάσαμε τα πάντα, δεν εξετάζουμε συγκεκριμένο... Είναι δύσκολο καλές μάλλον να επιμερίσει το κόστος, γιατί πολύ συχνά οι διακρίσεις βασίζονται σε προκαταλήψεις. Επομένως πάντα χρειάζεται ε, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση ε, ατόμων, που κοστίζει σημαντικά, συνολικά. Που εξηγεί, για παράδειγμα, γιατί δεν ασχοληθήκαμε και με την διάκριση για θρησκευτικού λόγους. Γενικά κόστε τώρα, λοιπόν όσον αφορά τη μεταγραφή του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Εθνικό Δίκαιο κτλ. Δεν εξετάσαμε το ζήτημα της παρακολούθησης, γιατί αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση με βάση την οδηγία. Είναι αποτελεσματικός τρόπος έτσι ώστε να υλοποιείται στην πράξη η νομοθεσία εθνικά, αλλά πάντως δεν είναι ε, κάτι που προβλέπεται στην οδηγία ως υποχρέωση του κράτους μέλους. Γι' αυτό δεν το αξιολογήσαμε. Πάντως, το κόστος ενός τέτοιου μηχανισμού εποπτείας είναι, μπορεί να είναι σημαντικό ανάλογα με τον τρόπο που θα ε, επιλεγεί. Δηλαδή, αν θα επιλεγεί η αυτορύθμιση ή αν θα δημιουργηθεί ένα σύστημα πιστοποίησης, ε, όπου, για παράδειγμα, θα απαιτείται από κάθε οργανισμό να, ε, να αποκτά ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τότε το κόστος αυξάνεται πολύ. Αυτά είναι λοιπόν παραδείγματα από τα κράτη-μέλη, στη Σουηδία είναι το μικρότερο κόστος, ε, το υψηλότερο ήταν στην Ισπανία. Βλέπετε στην οθόνη σας τα ποσά. Όμως, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα στοιχεία ε, είναι το αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων. Γιατί τα κράτη-μέλη έχουν στη διάθεσή τους πολλές επιλογές. Επομένως μπορεί να, τα ποσά να είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα ανάλογα με το τελικά πώς επιλέγει ένα κράτο μέλος να ποιες παραμέτρους επιλέγει ένα κράτο μέλος να λάβει ε, υπόψη του. Ίσως οι πιο σημαντικοί χώροι δράσης είναι αυτοί που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση σε κτίρια. Και εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες στα κτίρια όπου υπάρχει το κοινό και στα κτίρια όπου πηγαίνει κανείς στο, σε μια περιοχή όπου ζει κανείς στο σπίτι του μονάχα. Πρέπει να έχει πρόσβαση στο σπίτι του. Αν λάβουμε υπόψη λοιπόν αυτή την διαφορετική κατάσταση των δύο χώρων, έχουμε διαφορετικούς κανόνες για την πρόσβαση στα σπίτια. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για σπίτια τα οποία έχουν ιδιωτική ε, κατοχή και ιδιοκτησία και επομένω είναι διαφορετικά τα θέματα. Κοιτάξαμε τον αριθμό των κτηρίων, τι συνθήκες προσβασιμότητό του δεν ξεκινάμε φυσικά από μηδενική βάση, ξεκινάμε από περιοχές όπου υπάρχει ήδη προσβασιμότητα σε εμπορικούς χώρους, περίπου 40% είναι το ποσοστό αυτό, 10% για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες στα, σε κατοικίες. Υπάρχουν λοιπόν πάντα στοιχεία κατεκτήμηση. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που υπησέρχονται. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να τονίσω εδώ είναι ότι το κόστος θα εξαρτάται ε, επί τη βάση του τρόπου αλλαγών αν γίνεται μια αλλαγή ad hoc από ένα άτομο με αναπηρία ή αν γίνονται εκ των προτέρων αλλαγές για να διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρίες. Για τα εμπορικά κτίρια εδώ μπορεί να υπάρξει ένα κοινό δημόσιο πρότυπο. Υπάρχει μια νομική ασφάλεια με το να υπάρχουν εθνικά πρότυπα. Μια προσέγγιση λοιπόν ad hoc μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερο κόστος από ότι μια εκ των προτέρων συνολική ρύθμιση και αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον στον τομέα κατοικιών όπου τα άτομα αλλάζουν σπίτια μόνο παραδείγματος χάρη κάθε 20 χρόνια. Και Επομένω, ο αριθμό των ατόμων που χρειάζονται ειδική πρόσβαση στα 200 εκατομμύρια σπίτια που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περιορισμένο. Η άλλη διαφορά είναι να εφαρμοστεί μια τέτοια ρύθμιση μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 20 ετών ή σε ένα διάστημα μόνο 5 ετών. Αν είναι μεγαλύτερη χρονική περίοδος εφαρμογής, είναι μικρότερο το ετήσιο κόστος. Αν δούμε το κόστος αυτό σε ένα χρονικό ορίζοντα 100 ετών θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο να υπάρξει η μετασκευή όλων των κατοικιών. Αυτά είναι λοιπόν μερικά από τα κύρια συμπεράσματά μας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την δημογραφική αλλαγή στην κοινωνία μας, ότι εδώ το θέμα αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό, όσο γερνάει ο πληθυσμός, τόσο σημαντική είναι και η προσβασιμότητα σε όλα αυτά τα μέρη και έχουμε φυσικά μια μεγαλύτερη ε, ομάδα ανθρώπων και όχι μοναχά τα άτομα που έχουν αναπηρίες που ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν επισήμως αναγνωρισμένη <clears throat> αναπηρία αλλά έχουν δυσκολίες κινητικότητας ενδιαφέρονται για όλα αυτά. Ζωή στην τοπική κοινότητα τώρα. Κοίταξαμε και αυτό το θέμα γιατί και αυτό μας υποχρεώνει να το πράξουμε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών Και εδώ είναι το θέμα του τι πρέπει να γίνεται για να μεταφέρονται άτομα με αναπηρίες από θεσμικά ιδρύματα στην κοινότητα όπου ζουν. Εδώ είναι ακόμα περισσότερες οι παράμετροι και έχουμε πολύ μεγαλύτερα περιθώρια παραγωγής χάρη για την περίοδο εφαρμογής 5 ετών. Έχουμε 269 μέχρι 250 εκατομμύρια για τη Ρουμανία για να γίνει η μεταφορά από θεσμική περίθαλψη σε μια κοινότητα η οποία ε, παρέχει την περίθαλψη. Δεν θεωρούμε ότι είναι εφικτό να περάσουμε απόλυτα από ένα θεσμικό σύστημα περίθαλψης σε ένα σύστημα περιθάλψης από την τοπική κοινότητα. Αυτό θα σημάνει ότι πρέπει να παραμείνει ένα διτό σύστημα το οποίο αυξάνει το κόστος. Βλέπετε τώρα ότι η Σουηδία δεν έχει καθόλου θεσμικά ιδρύματα. Όλη η περίθαλψη γίνεται σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και αυτό μπορεί να είναι ένας απότερος στόχος, πρέπει να λάβει υπόψη όμως ότι το κόστος είναι περίπου διπλάσιο το κόστος σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος και πιστεύω ότι αυτό θα το δείτε όσο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα για την εφαρμογή, το χαμηλότερο το ετήσιο κόστος. Πάμε τώρα στα μέσα ενημέρωσης. Εδώ δεν υπάρχει ιδιαίτερη σαφήνεια για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό. Μπορεί παραγωγικά να ζητηθεί από όλα τα κανάλια να βάζουν υποτίτλους στις εκπομπές τους. Εμείς κοιτάμε κυρίως να βρούμε μια πιο αναλογική προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη και τις ενέργειες που κάνουν τα κράτη-μέλη. Είδαμε το κόστος λοιπόν για τη, τα μεγαλύτερα κανάλια. Προσπαθούμε να επιτύχουμε μια παροχή υποτίτλων για τα περισσότερα άτομα με αναπηρία. Ε, 100% λοιπόν υποτιτλισμό για τα μεγαλύτερα κανάλια. Βλέπετε ότι το κόστος είναι πολύ μεγάλο. 1,9 εκατομμύρια 1.900 εκατομμύρια μάλλον για τα κράτη-μέλη και φυσικά έχει να κάνει και με το χρόνο ε, εκπομπής και για την ε, ε, εφαρμογή που γίνεται. Τέλος, έχουμε δύο ακόμα περιοχές που εξετάσαμε για τη διάκριση βασιλικίας. Η διάκριση βασιλικίας ήταν ένας πολύπλοκος τομέας. Για τον τομέα της υγείας μιλάμε για ένα οικονομικό τομέα ο οποίος καλύπτει δισεκατομμύρια ευρώ Δεν ξέρουμε λοιπόν αν η ίση μεταχείριση αποτελεί μια μορφή διάκρισης γιατί έχουμε ηλικιωμένα άτομα τα οποία παίρνουν μια ε, αντιμετώπιση διαφορετική από αυτή των νέων αλλά εδώ πέρα φυσικά υπάρχουν ανάγκες διαφορετικές. Φαίνεται ότι υπάρχουν ε, στοιχεία διακρίσεων τα οποία επηρεάζουν πολλούς ε, ασθενείς. Και βεβαίως το θέμα είναι και τι μέθοδος θεραπείας χρησιμοποιείται και αν έχουν συγκατατεθεί ή όχι. Είναι λοιπόν διαφορετικά τα πράγματα αν κάνει κανείς χημιοθεραπεία, αν υπάρχει μεταμόσχευση. Είναι λιγότερες πιθανότητες για τους άνω των 65 να λάβουν ε, μόσχευμα Αλλά είναι δύσκολο να πούμε αν αυτό είναι ένα παράγον διακριτική μεταχείριση ή όχι. Πάντω, βλέπετε ότι το κόστο διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην δημοκρατία τη Τσεχία δίδονται κάποια ωφέλη, ενώ στην Γερμανία δεν υπάρχει κανένα όφελο, Πρόκειται λοιπόν για μια αποτίμηση που είναι διαφορετική ανατομέα και αναχώρα. Τα πράγματα αλλάζουν ως προς την κατάθλιψη. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για την ε, ψυχολογική υγεία και για τους άνω των 65. Όταν δεν ε, είναι αντικείμενο θεραπείας, είναι και λόγος αυτοκτονιών για τους άνω των 65. 10% λιγότεροι από οι νεότεροι άνω των 65 ε, έχουν διάγνωση και λαμβάνουν ε, φαρμακευτική περίθαλψη για την κατάθλιψη. Είδαμε όμως ότι αν υπήρχε η θεραπεία με τη διάγνωση θα υπήρχε και ένα σαφές κέρδος για όλα τα κάτι μέλη. Θα υπήρχε μεγαλύτερη η άνεση να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί στη δουλειά τους και βεβαίως και αυτό θα ήταν και ένα τομέας, ένα παράγων ίσης μεταχείρισης. Ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό, το βασικό ή ενδεχόμενο κόστος που μας απασχόλησε είχε να κάνει με το κατά πόσον υπάρχει ίση μεταχείριση ως προς το φορολογικά ε, ως προς τις ε, φορολογικές ελαφρύνσεις. Υπάρχουν ε, για τα παντρεμένα ζευγάρια τέτοιες ελαφρύνσεις αλλά μόνο ένα στα πέντε κράτη-μέλη είτε δεν είχε καμία νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, είτε και προέβλεπε τη δυνατότητα ομόφυλων ε, ε, συντρόφων ή ομοφυλόφιλους γάμους. Ο αριθμός πάντως εταιρικών, ε, των συμφώνων συμβίωσης στις χώρες που κοιτάξαμε είναι πολύ χαμηλός για τους ε, ομόφυλους. υπάρχει λοιπόν ανάγκη να είναι ίση μεταχείριση και ως προς τους φόρους, διότι είναι τόσο λίγοι άνθρωποι που καλύπτει αυτή η κατηγορία που το κόστος θα ήταν πάρα πολύ μικρό. Τα συνολικά μας τώρα πορίσματα. Σε όλο το φάσμα των θεμάτων που μας απασχόλησαν, στις περισσότερες περιοχές το κόστος δεν θα ήταν σοβαρό. Μιλάμε για πολύ συγκεκριμένους τομείς, οπότε η υλοποίηση της οδηγίας στους περισσότερους τομείς δεν θα προκαλούσε μεγάλο κόστος. Εκεί που θα προκαλούσε μεγάλο κόστος είναι στην αντιμετώπιση της διακριτικής μεταχείρισης και την πρόσβαση στις υποδομές. Εκεί φαίνεται ότι το κόστος αυξάνεται γεωμετρικά και σε ό,τι αφορά τη ρυθμιστική συμμόρφωση και εκεί το κόστος είναι σχετικά χαμηλό. Βέβαια, όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος για συμμόρφωση με την υλοποίηση της οδηγίας, τόσο μικρότερο θα είναι και το κόστος. Εδώ όμω απαιτείται και κάποια ισορροπία, διότι η συμμεταχείριση είναι θεμελιώδης δικαίωμα. Ε, δικαίωμα, οπότε η σωστή ισορροπία μεταξύ του χρόνου θα το πετύχει κανείς αυτό και του κόστους είναι σημαντικός παράγον. Και όπως έλεγα και προηγουμένως υπάρχει μια σειρά από επιλογές υλοποίησης που προσφέρονται στα κάτι μέλη. Από την πιο ε, συνολική μέχρι την εξελαχίστων προσέγγιση. Ε, προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε και στον υπόλοιπο κόσμο ποια θα ήταν η πιο λογική προσέγγιση. Αυτά ήταν τα πορίσματά μας ως τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση της μελέτης. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα. Κύριε Ρωμέβα, δεν ήσασταν εδώ όταν ε, ανέφερα ότι επί χρόνια, επί σειρά ετών, μπλοκάρει το Συμβούλιο ε, και σέρνεται προκειμένου να μην εξετάζει την οδηγία για την ίση μεταχείριση. Είναι πραγματικά δυσάρεστο αυτό, είναι πολιτικό θέμα και καλούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, πάρει σοβαρά ε, το θέμα αυτό. Ήδη απευθυνθήκαμε και στους υψηλόβαθμους ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον ίδιο τον Πρόεδρο Μπαρόζο, και όμως η ιστορία αυτή δεν έχει τελειώσει. Θέλουμε λοιπόν εδώ να ακουστεί ότι χωρίς ίση μεταχείριση ενώπιον του νόμου ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχουμε κρίση μόνο του ευρώ και της οικονομικής διαχείρισης. Εμείς ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών, εκλεγμένοι εκπρόσωποι, θα είμαστε σε κρίση μέχρι το θέμα αυτό να παραμένει ανεπιλήτο. Κύριε Ρωμέβα, ας ακούσουμε τώρα τι έχετε να μας πείτε ως εισηγητής για την οριζόντια αυτή οδηγία για την ίση Και μετά θα ανοίξει η συζήτηση. I have also the, is the Commission Ευχαριστώ, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, θα δώσετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ελληνική Προεδρία. Μήπως θα ήταν καλύτερα να μιλήσει πρώτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκληθεί και η Ελληνική Προεδρία και η επερχόμενη Ιταλική Προεδρία ε, έχουν εκπροσώπους εδώ και θα έχουν τη δυνατότητα να ε, μιλήσουν. Έχετε τώρα το λόγο εσείς όμως. Ωραία, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να βάλουμε ένα πλαίσιο σε αυτή τη συζήτηση γιατί πράγματι είναι μια συζήτηση η οποία έχει διαρκέσει πολλά χρόνια. Όταν, όταν ξεκινήσε τη θητεία του αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα από τα ζητήματα προσπάθησε να θέσει ήταν να δημιουργηθεί μια πολιτική όθηση έτσι ώστε αυτή η οδηγία να προχωρήσει. Γνωρίζουμε ότι το μπλοκάρισμα ήταν στο Συμβούλιο, η Επιτροπή έκανε τη δουλειά της. Το λόγος που είναι μπλοκαρισμένη αυτή η οδηγία είναι βασικά γιατί κάποιες κυβερνήσεις αντιτίθενται σε αυτήν για διάφορους λόγους. Κάποιες ανοιχτά, άλλες όχι. Και αυτό το θεωρώ όχι απλώ λυπηρό, αλλά επίσης ένα απαράδεκτο μήνυμα από δημοκρατική απόψεως στους Ευρωπαίου πολίτες. Προσπαθήσαμε λοιπόν να συνεργαστούμε πολύ στενά με τι προεδρίες. ορισμένε από αυτές ε, εργάστηκαν ε, ενεργά. Στην αρχή ε, εργαστήκαμε για παράδειγμα πολύ καλά με την Ισπανική και μετά τη Βελγική Προεδρία. Με εκείνες τις δύο προεδρίες είχαμε πολύ καλή συνεργασία, αλλά Σύντομα διαπιστώσαμε και αντιληφθήκαμε ότι αυτές οι συζητήσεις θα είναι πολύ δύσκολες. Στο Συμβούλιο, ενώ τι συζητήσει στο Συμβούλιο, όχι στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο, α μην ξεχνάμε ότι είχε ήδη εγκρίνει το κείμενο, είχε ε, λάβει θέση στην προηγούμενη θετία του, η οποία συνεχίζει να ισχύει μια και δεν την τροποποίησε. Άρα η θέση του Κοινοβουλίου ήταν ε, ξεκάθαρη. Είναι ξεκάθαρο επίση ότι το μπλοκάρισμα προκύπτει στο Συμβούλιο η μία Προεδρία μετά την άλλη προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να προχωρήσει το θέμα. Γνωρίζω ότι στο τεχνικό επίπεδο ε, εκεί τα πράγματα έχουν ξεκαθαριστεί, Οι όποιες ανησυχίες έχουν ε, διευκρινιστεί. Επομένως το πρόβλημα που παραμένει είναι πολιτικό, δεν είναι τεχνικό. Και γι' αυτό γνωρίζουμε ότι δεν είναι το πρόβλημα εύκολο να λυθεί. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι ίσως ένα από τα ζητήματα που αποσχολεί τα κράτη-μέλη να είναι το κόστος τη εφαρμογή της οδηγία. και γι' αυτό ίσως θα ήταν σκόπιμο να εκτιμήσουμε αυτό το κόστος. Τι, σημαίνει, τι θα σημάνει μάλλον η υλοποίηση αυτή τη οδηγία. Θα είναι τόσο ακριβή. Όπω είπατε, δεν έχει σχέση το πώ θα ορίσουμε το κόστο με, με, με, τα, με τα δικαιώματα και θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό όχι μόνο για τους πράσινους, αλλά φαντάζομαι και με τους άλλους συναδέλφους, τους περισσότερους με τους οποίους συνομιλώ, η αρχή της ισότητας οφείλει να γίνεται σεβαστή ανεξαρτήτως από το κόστος. Η ισότητα των δικαιωμάτων είναι απείρως πιο σημαντική από την οικονομική διάσταση του θέματος. Ωστόσο, μιας και υπήρχε αυτή το, το μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο, είπαμε ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον να αξιολογήσουμε και την οικονομική παράμετρο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μονάδα αξιολόγηση αντικτύπου που μα έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή μα. Μετά ε, ζητήσαμε την αρρωγή τη ε, εταιρεία Μιλιό και άλλων για να γίνει αυτή η μελέτη. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω κάποια πράγματα για τη μελέτη και τα συμπεράσματά τη. Όσον αφορά την ίδια τη μελέτη, Γνωρίζουμε και μας απασχολούσε από την αρχή ότι αυτό που του ζητήσαμε ήταν τιτάνιο έργο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πρώτα απ' όλα να οριοθετήσει κανείς το θέμα. Και σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζεται απλώς να βασιστεί σε εκτιμήσεις. Είναι πολύ δύσκολο συγκεκριμένα να αξιολογήσει κανείς, να εκτιμήσει μάλλον κανείς ποιο θα, ποιο θα είναι το κόστος. Αλλά και αυτό είναι χρήσιμο για να αντιταχθούμε στα κράτη-μέλη εκείνα που ε, αναφέρουν συχνά το επιχείρημα όχι αυτό το, αυτές οι επιλογές, αυτές οι ε, πολιτικές θα είναι πολύ ε, ακριβές, θα, θα κοστίσουν πολύ, γιατί το ζήτημα θα έπρεπε να τίθεται με πολιτικούς όρους και όχι με οικονομικούς όρους. Σε όλους τους τομείς που εξετάζουμε, από ε, όλους αυτούς τους τομείς μάλλον μπορούμε να επιλέξουμε έναν στον οποίο θα μπορούσε κανείς να λάβει υπόψη του και το ζήτημα του κόστους και είναι το ζήτημα των ατόμων με αναπηρία. Για τους υπόλοιπους τομείς θα έλεγα ε, αν όχι ότι είναι άσχετο το ζήτημα και δεν πρέπει να το συζητάμε, εν πάση περιπτώσει εάν υπάρχει πρόβλημα μπορούν να βρεθούν αντισταθμιστικά μέτρα ή άλλες προβλέψεις στο πλαίσιο της οδηγίας. Χαίρομαι λοιπόν που η εκθέση ε, ξεκαθαρίζει αυτές τις έννοιες. Επίσης να πω ότι όταν αρχίζουμε να συζητάμε για το κόστος, θα πρέπει να μην ξεχνάμε και το όφελος. Το όφελος που θα έχει η υλοποίηση αυτής της οδηγίας. Το να έχει κανείς μια ε, καταρχήν πολιτική κατά των διακρίσεων σε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό καταπολεμά συνολικά τις διακρίσεις και μειώνει το κόστος που προκαλούν οι ίδιες οι διακρίσεις, ας πούμε. Μπορούμε λοιπόν να δούμε και το ζήτημα από την πλευρά του ωφέλους που θα, θα υπάρξει. Και τέλος, υπάρχει ένα συμπέρασμα πολύ ξεκάθαρο από αυτή την μελέτη, ότι τα κόστη αυτά που εξετάστηκαν, δηλαδή εκείνα που προέρχονται από διακρίσεις με βάση, προκαταλήψ, βάση προκαταλήψεων, αυτά τα κόστη δεν πρόκειται να είναι σημαντικά. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί ενώ σε κάποιους τομείς προφανώς θα υπάρχει κόστος, το συνολικό τελικό αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να το εξετάζουμε με οικονομικού όρους, να μην το δούμε δηλαδή με βάση το αν κοστίζει πολύ ή λίγο. Αυτό μας δίνει τώρα τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Διαφέρει εάν η οδηγία χρειαστεί να υλοποιηθεί σε 5-10 χρόνια. Αυτό είναι κάτι το χρονοδιαγραμμα υλοποίηση. διαφερει εαν προσπαθήσαμε να περάσουμε και στις κυβερνήσεις που κολυσεργούν και δεν επιθυμούν τη συζήτηση του θέματος. Είναι λοιπόν σημαντικό να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. δεν το λέω μόνο ως ε, πρώην, μάλλον μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί δεν πρόκειται να ξαναθέσω υποψηφιότητα. Το λέω για τους επόμενους. Στην επόμενη θητεία, πολύ θα ήθελα να είναι ένα από τα επόμενα ζητήματα που θα προωθηθούν στην επόμενη θητεία, αλλά δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξο, τουλάχιστον στο βράχι, βραχυπρόθεσμα. Γι' αυτό λοιπόν πολύ θα ήθελα να δω η ελληνική και η ιταλική προεδρία να το λάβουν αυτό το ζήτημα σοβαρά υπόψη τους και να το προωθήσουν στο Συμβούλιο. Σα το ζητώ, αλλά σας ζητώ να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό με τρόπο πολιτικά υπεύθυνο και κάποια σύντομα σχόλια, μάλλον ένα τελευταίο σχόλιο για το περιεχόμενο της έκθεσης. Σε ορισμένα σημεία δίνει την εντύπωση ότι κάποιες δράσεις μπορεί να είναι πολύ ακριβές. Αλλά σε ορισμένα από τα παραδείγματα που δίνονται μέσα στην έκθεση, τα παραδείγματα αυτά δεν συνδέονται άμεσα με την οδηγία. Αν δηλαδή δούμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, η ίδια η υλοποίηση της οδηγίας δεν θα είχε επιπλέον κόστος. Με όλα αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ θα ήθελα να ακούσω και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δύο Προεδριών, της Ελληνικής και της ελληνική Προεδρίας και φυσικά τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρωμέβα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει σχόλια. Εάν όχι, στρεφόμεθα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Άλβαρο Ολιβέρα θέλει να λάβει το λόγο. Ο κύριος Στάιν, θέλετε να πείτε κάτι, παρακαλώ. Λέγομαι Στάιν, είμαι επικεφαλής της ομάδας ίσης μεταχείρισης στην Γενική Διεύθυνση για τα θέματα δικαιοσύνη. Εμεί έχουμε διαπραγματευτεί λοιπόν αυτή την οδηγία και την έχουμε φέρει στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το να τονίσω απερίφραστα και απλά ότι είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι προς την πρόταση αυτή. Δεν υπήρξε ποτέ καμία η παραμικρή αμφιβολία ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στο Συμβούλιο που όπως ξέρετε χρειαζόμαστε ομοφωνία για να εγκριθεί αυτή η πρόταση, η Κομισιόν δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει αυτή την πρόταση, την προωθεί με κάθε ευκαιρία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε και συμμαχίες που θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο Συμβούλιο και να, να έχουμε μια γενική υποστήριξη. Έχουμε επιτύχει πολλά λοιπόν τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, αλλά δεν είμαστε και τόσο απεσιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή σε σχετικά λογικό χρονικό διάστημα του πολιτικού κλίμα. Ίσως είμαι υπεραισιόδοξο, αλλά συνεχίζουμε την προσπάθειά μα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την υποστήριξη που πήραμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω από την εισηγητή για το θέμα αυτό, το Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει με απόλυτη επιμονή και χωρίς υπαναχώρηση το θέμα αυτό και έχει ζητήσει από το Συμβούλιο να μην αδρανεί για το θέμα αυτό, αλλά να συνεχίσει την επεξεργασία του. Και πιστεύω ότι αυτή η πίεση εξηγεί σε κάποιο βαθμό, γιατί το Συμβούλιο εξακολουθεί να ασχολείται με το θέμα αυτό, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική ε, συνένεση στο Συμβούλιο για τα θέματα αυτά. Κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη του να το θέσει στο αρχείο τη στιγμή που υπάρχει τέτοια υποστήριξη από το Κοινοβούλιο και επίσης και από το μεγαλύτερο μέρος των κρατών μελών απλώς δεν μπορούμε να πετύχουμε την απαραίτητη ομοφωνία η οποία χρειάζεται. Χαιρόμαστε λοιπόν για την υποστήριξή σας και είδα ότι η τελευταία ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό ήταν πέρσι το καλοκαίρι που ήταν η πέμπτη επέτειος της ε, υποβολής αυτής της πρότασης και το Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να τονίσει ότι θέλει να συνεχίσει να την υποστηρίζει. Βρισκόμαστε λοιπόν σε, στην ίδια κατεύθυνση με το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Συζητάμε σήμερα την, την ε, <clears throat> συμπληρωματική έκθεση αντικτύπου που έγινε από τον Φορέα Μιλίο. Θέλω να πω ότι κατανοώ ότι αυτή η μελέτη είναι ένας τρόπος να κρατήσουμε ζωντανή τη συζήτηση και μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη ε, βάση για να προωθήσουμε επιπλέον την έγκριση αυτής της πρότασης. Επειδή η Κομισιόν είναι το όργανο το οποίο είναι αρμόδιο για να παρουσιάσει μια πλήρη έκθεση αντικτύπου με όλες τις πτυχές που εμπλέκονται σε όλες τις πολιτικές. Κατανοώ πόσο μεγάλες είναι οι δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως Επιτροπή για να φέρουμε σε πέρα σε αυτό το εγχείρημα. Έχουμε συνεργαστεί με το Μιλίο. Έχουμε δώσει πληροφορίες επί τη βάση της δικής μας για την δική μας έκθεση αντικτύπου κατανοούμε το πόσο σημαντική προσπάθεια έχει γίνει από την πλευρά τους για να μπορέσει να φέρει σε φω νέα στοιχεία και νέες αξιολογήσει για το κόστος και το όφελος. Δεν μπορώ τώρα να μπω σε λεπτομέρειες για συγκεκριμένε θέσει που έχει αναφέρει η έκθεση αντικτύπου της Μίλιο Πιστεύω όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συμβολή και θέλω να τονίσω αυτό που είπε ο εισηγητής προηγουμένως, ότι όταν μιλάμε για δυνητικά σημαντικό κόστος, μιλάμε πάντα για ένα πολύ περιορισμένο τμήμα της οδηγίας εν γέννη. Το πρώτο συμπέρασμα λοιπόν της έκθεσης αντικτή που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι για το μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής αυτής της οδηγίας δεν θα προκύψει συνολικό σημαντικό κόστος το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα αντεπιχείρημα κατά <clears throat> αυτής της οδηγίας και της πρότασης. Μιλάμε για μονάχα συγκεκριμένους τομείς όπου θα υπάρξει πρόσθετο κόστος και φυσικά τα θέματα της ε, κατάλληλη στέγαση για τα άτομα με αναπηρία είναι ο χώρος όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικό κόστος. Αλλά, και εδώ θέλω να κάνω αυτό το γενικό σχόλιο, έχοντας κάποια εμπειρία με τις εκθέσεις αντικτύπου και επιπτώσεων, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει <clears throat> κάποια εγγενής μεροληψία σε μια τέτοια έκθεση, χωρίς δεν υπάρχει καμία πρόθεση, ώστε να προσπαθεί να δει κανείς την οικονομική μοναχαπτυχή <clears throat> για τα θέματα αυτά, είναι πάντα πολύ πιο εύκολο να περιγράψει το κόστος κανείς παρά το όφελος. Γιατί το κόστος είναι άμεσο κόστος, πόσο χρειάζεται δηλαδή για να εφαρμοστεί ένα <clears throat> μέτρο, ενώ τα ωφέλη είναι έμεσα και άδειλα και δεν είναι τόσο εύκολο να τα, προσμε... να τα καταμετρήσει κανείς. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση να υπερεκτιμά κανείς το κόστος έναντι του ωφέλους και υπάρχει ένα πρόσθετο στοιχείο, το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό στα πλαίσια αυτής της οδηγίας, ότι συγκεκριμένα το κόστος και το όφελος με τον τρόπο που κάνουμε εμείς την αξιολόγησή μας στην Κομισιόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε οικονομικό επίπεδο. Αυτό είναι μία πτυχή του κόστους και του ωφέλους που είναι σημαντικό στην ανάλυση, αλλά εμείς θα πρέπει να δούμε και το κοινωνικό κόστος και το κοινωνικό όφελος το οποίο μπορεί να προκύψει και όχι μονάχα το οικονομικό κόστος και τα οικονομικά ωφέλη. Σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση είναι προφανές ότι το κοινωνικό κόστος της έλλειψης ενός πλαισίου <clears throat> ίσης μεταχείρισης και η αποστέρηση από τα κοινωνικά ωφέλη μιας τέτοιας ρύθμισης είναι πάρα πολύ σημαντικά και επομένως πρέπει να παίξουν κάποιο ρόλο να καταμετρηθούν στην πλάστιγκα. Κύριε Στάινερ, έχουμε χρονικό πρόβλημα. Έπρεπε να είχαμε τελειώσει στις 12 ε, και έχουμε άλλο ένα σημείο. Σας παρακαλώ λοιπόν πώς πατήστε να συνοψίσετε. θα είμαι σύντομο. Το δεύτερο θέμα λοιπόν που οδηγεί σε κάποιες στρεβλώσεις στην, ε, όπως είπα υπάρχει το στοιχείο της υπερεκπροσώπησης του οικονομικού στοιχείου και υποεκπροσώπησης του κοινωνικού κόστους και ωφέλους γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να ποσοτικοποιηθεί το πρώτο και υπάρχει γενική τάση για την ποσοτικοποίηση. Ένα δεύτερο γενικό σχόλιο το οποίο όμως θα ήθελα να κάνω για τα θέματα αυτά είναι ότι πρέπει να βρει κανείς το σωστό σημείο αναφοράς. Η έκθεση αντικτύπου και επιπτώσεων προσπαθεί να αναλύσει τα ωφέλη και το κόστος σε σχέση με το τωρινό σημείο, με το status quo. Τι θα μπορούσε να προκύψει ως κόστος και όφελος. Εδώ όμω υπάρχει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας και θα παραμείνω μόνο σε αυτό το σημείο το οποίο όμω νομίζω ότι είναι μεγάλη σημασία. Πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ήδη μία νομοθετική υποχρέωση ιδιαίτερα για τον τομέα όπου το μιλίο βρήκε να υπάρχει το μεγαλύτερο δυνητικό κόστος που είναι ο τομέας της, ε, των ατόμων με αναπηρία. Έχουμε τη σύμβαση του ΟΗΕ που δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύει όλα μας τα κράτη. Από τα συμπεράσματα που βρίσκονται στην ε, σύνοψη για τους λήπτες αποφάσεων της έκθεσής μας, λέει η Μιλία ότι εφόσον όλα τα κατημέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση αυτή θα μπορούσε κανείς να θεωρεί ότι το κόστος το οποίο θα προκύψει από την εφαρμογή των μέτρων για τους αναπήρους προκύπτει καταρχήν από τις υποχρεώσεις που έχουν συναυθεί με την υπογραφή και την κύρωση της, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Επομένως το κόστος που υπολογίζει η Μιλιέ δεν είναι το πραγματικό κόστος λήψης των μέτρων αυτών, γιατί κάποια μέτρα είναι ήδη υποχρεωτικά επί τη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Αν, αν πάρουμε λοιπόν το σωστό σημείο αναφοράς για αυτή την οδηγία, όταν θέλουμε να υπολογίσουμε το πραγματικό κόστος της οδηγίας, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τι αναπηρίες είναι στοιχεία που αποτελούν ήδη συμβατικέ υποχρεώσει τη ευρωπαικη ενωση επομενω η οδηγία θα έχει ένα πολύ μικρό πρόσθετο κόστο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη όταν συγγίζουμε τα υπέρ και τα κατά της εφαρμογή αυτής τη συγκεκριμένης πρόταση. Και κατά τα άλλα νομίζω ότι ο εισηγητής έχει ήδη κάνει κάποια σχόλια τα οποία θα έκανα και εγώ ότι σε ορισμένου ε, τομεί ξεπερνάμε ήδη το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία όταν μιλάμε, παραδείγματο χάρη, για τα φορολογικά πλεονεκτήματα. Αυτά είναι εκτό του πλαισίου τη οδηγία ή όταν μιλάει για πρόσβαση σε δημόσιου δρόμου, λεωφόρου. Κλείνω λοιπόν λέγοντα να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει ήδη δέσμευση από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το πώς υποεκτιμούνται τα κοινωνικά ωφέλη. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα η ελληνική προεδρία. Θέλετε να πάρετε το λόγο για πολύ λίγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς να χαιρετήσω τη συνάντηση που διοργανώσατε σήμερα Νομίζω ότι θα συμβάλλει στο να έχουμε μια καλύτερη προβολή του θέματος και να διασκεδάσουμε κάποιες παλιές ανησυχίες που απομένουν στο επίπεδο του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Από τότε που υποβλήθηκε αυτή η πρόταση οδηγίας, ξέρετε ότι η Ελλάδα είχε θέση μάλλον θετική και δημιουργική για την εξέλιξη του όλου θέματος. Και σε αυτό το πλαίσιο ξεκινήσαμε τις συζητήσεις στην ομάδα εργασίας στις αρχές Μαρτίου. Ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Συμμερίζομαι απολύτω την ανάλυση περί κόστους ε, και τις παρατηρήσεις που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τον ε, εισηγητή για το κόστος. Απλώς να θυμίσω, επειδή εργάστηκα ως αρχιτέκτονας επί 30 χρόνια για τα θέματα της πρόσβασης, δεν πρέπει να μετρήσουμε μόνο το άμεσο κόστος, πρέπει να προσπαθήσουμε να μετρήσουμε και τα ωφέλη, το ε, έμεσο κέρδος μέσω αυτών των ε, προσαρμογών, των πολεοδομικών. Μην ξεχνάμε ότι μια πολεοδομική αλλαγή, είτε αφορά την πρόσβαση, είτε τον δημόσιο ιδιωτικό χώρο, θα επιτρέψει την πρόσβαση των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας. Θα συμμετέχουν στο κοινωνικό βίο, στην ζωή της κοινωνίας. Και θα υπάρξουν συνέπειες σορευτικές, θετικές σορευτικές συνέπειες που δύσκολο είναι να τις υπολογίσουμε. Πάντως, να σας καθησυχάσω ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται για το θέμα αυτό. Μας απασχολεί και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσει. Ευχαριστούμε για τις ε, σας. Να επιστρέψουμε στο Προεδρείο. Κύριε Άιτεν, θέλετε να παρέμβετε ο κύριος Μόλτερ. Και μετά θα ακούσουμε τον εισηγητή μας. Δεν γνώριζα αυτό το θέμα πολύ καλά από προηγουμένω, αλλά άκουσα μεγάλο ενδιαφέρον, ιδίω τόσο είπε ο να τον συγχαρώ για την αφοσίωσή του μάλιστα επί του θέματος. Οι εξηγήσει που μας έδωσαν ήταν πολύ διαφορετικές για μένα. Μια ερώτηση τώρα. Υπάρχει ένα κατοσμέλο, η Γερμανία, που δυσκολεύεται με την υλοποίηση της οδηγίας αυτής. Μου λέτε τι έχει γίνει ως τώρα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμμερίζομαι την την βάθος ανάλυση που θα χρειαστεί, γιατί το τελικό συμπέρασμα είναι ότι το κόστος του να υλοποιηθεί αυτή η οδηγία θα πρέπει να συγκριθεί με το ενδεχόμενο κόστος του να μην υλοποιηθεί. Και συμφωνώ απολύτως ότι το κέρδος είναι λιγότερο εύκολο να καταμετρηθεί από το κόστος, διότι ε, μπορεί να εντοπίζονται σε μεγαλύτερο φάσμα χρόνου. Οπότε ελιθεύει αυτό. Χαίρομαι που και το Συμβούλιο συμμερίζεται αυτή την άποψη. Και όσο για την κατάσταση στη Γερμανία, να πω ότι το παράδοξο είναι ότι η κυβέρνηση της Γερμανίας είναι από τις πιο προσφυλακτικές το να ισχύσει η οδηγία αυτή. Αλλά τα περισσότερα που προβλέπει η οδηγία ούτως ή άλλως ισχύουν ε, στη Γερμανία και προβλέπονται. Είναι καλυμμένοι οι Γερμανοί. Αυτό είναι το πλέον παράδοξο. Πάντως ε, ελπίζουμε ότι με την αλλαγή της κυβέρνησης ε, θα έχουμε κάποιο περιθώριο λεγμών και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποια μετατόπιση Στι απόψεις τη Γερμανία Και χαίρομαι και για την αισιοδοξία τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το θέμα αυτό. Διότι η τωρινή ή η μελλοντική Προεδρία ελπίζουμε να θέσουν το θέμα αυτό επιτάπητο για να εξεταστεί. Υπό αυτήν την έννοια να πω ότι λυπούμε που δεν θα είμαι αυτός ο οποίος θα ε, οδηγήσει σε αίσιο πέρας το δοσχέ αυτό, όμως με μεγάλη χαρά θα έρθω όταν γίνει αυτό για να γιορτάσω μαζί σας και με όλους τους πολίτες αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε λοιπόν για τη μελέτη και όλους τους συναδέλφους για τη δουλειά τους ως τώρα και βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο εδώ στην επίλυση όχι μόνο τεχνικών προβλημάτων, αλλά στη διευκόλυνση των συζητήσεων, διότι οι προεδρείς εναλλάσσονταν, όμως η Επιτροπή ήταν πάντα παρούσα. Απαντώντα σε όλες τις ερωτήσεις που ενδεχομένω είχαμε. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε και καλό είναι να το να ακουστεί. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ και ελπίζω σύντομα να έρθουμε και να πούμε διαφορετικά πράγματα από αυτά που είπαμε σήμερα. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλα σχόλια. Έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο μας και πλησιάζουμε το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Έχουμε ένα ακόμα σημείο για πληροφόρηση. Κύριε Μούλτερ, για την αντιπροσωπεία μας στην Βαλέτα, στη Μάλτα, για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης του Ασύλου. Έχετε το λόγο για να κάνετε την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Τρεις βουλευτές πήγανε στο γραφείο του ΕΑΣΟ στη Μάλτα. Υπήρξε πολύ καλή υποδοχή. Πήραμε πλήρη πληροφόρηση για τις λειτουργίες του κέντρου. Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους των κρατών μελών. Πληροφορηθήκαμε για την κατάσταση των προσφύγων στην Μάλτα, που είναι μια μικρή χώρα που υφίσταται τεράστια πίεση από τον αριθμό των προσφύγων. Συζητήσαμε με το κοινό, κάναμε μια βραδινή συνάντηση με ανθρώπους από τον τοπικό πληθυσμό και αυτούς που έχουν πάρει το δικαίωμα του ασύλου και η γενική μας εντύπωση είναι ότι είναι όλο και πιο σημαντικός ο ρόλος του, του γραφείου για τη συλλογή πληροφοριών και για την κατάρτιση και δείχνει την αξία του ιδίως σε μια στιγμή που υπάρχει μεγάλο ρεύμα προσφύγων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Η κυρία Μετσόλα θέλει να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μούλτερ γιατί υπήρξε επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας με υποδειγματικό τρόπο. Ήταν τιμή για μένα να μεταβώ στη χώρα μου με αυτή την πρώτη αποστολή που, στην οποία συμμετέσχα μετά την εκλογή μου και φυσικά υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την κατάσταση μετανάστευσης και ασύλου στη Μάλτα και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους ενός φορέα που έχει σαν κεντρικό στόχο του να υποστηρίξει τη διαδικασία παροχής ασύλου και την ε, επανεγκατάσταση των ε, προστατευόμενων από άσυλο από το ένα κράτος σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζητήσαμε όλοι για το πώς μπορεί το γραφείο αυτό να βοηθήσει τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ένα δυσανάλογο βάρος ετούν των ασύλου και πώς θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια πιο ισοδίκια κατανομή των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών για το τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Ο κύριος Ντεμπλάζη, η κυρία Γκυγιόμ, ο κύριος Μπρόντς. Θέλετε κύριε Μπρόντς, έχετε το λόγο. Ένα ερώτημα μονάχα. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε για τα, τις ομάδες ατόμων που συναντήσατε. Ήταν άτομα τα οποία είχαν άμεση εμπλοκή στα θέματα αυτά, τα, αυτοί οι οποίοι ζητούσαν άσυλο ή μέλη τοπικών οργανισμών, αλλά μιλήσατε και σε απλούς ανθρώπους και τι πιστεύανε για όλα αυτά. Κύριε θέλετε να πείτε κάτι κι εσείς. Να προσθέσω μονάχα ότι σε σχέση με αυτά που αναφέρθηκαν, προφανώς το γραφείο για την υποστήριξη του, της παροχής ασύλου είχε ένα αποτελεσματικό και αποφασιστικό ρόλο για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν μεγάλες πιέσεις σε ό,τι αφορά τους ετούντες ασύλου. Πρέπει να τονίσουμε όμως επίσης ότι στην αποστολή αυτή του Γραφείου για την Υποστήριξη του Ασύλου υπάρχει και ο ρόλος να υποστηρίξει μια μακροχρόνια αναζήτηση, υποστήριξη το Συμβούλιο για μια πιο μακροχρόνια πολιτική και μια υποστήριξη προς την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων όταν ανακύπτουν. Στη Μάλτα υπάρχει μια ιδιαίτερη πίεση και εκεί πέρα παίζει και το ρόλο του το γραφείο αυτό για να βρεθεί μια λύση και επίσης καλείται το γραφείο αυτό να δώσει υποστήριξη σε εγκάρσιο θα έλεγα επίπεδο για όλες τις πολιτικές ασύλου. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ε, ενήμεροι για όλα αυτά τα θέματα και το ρόλο που παίζει το γραφείο. Ευχαριστώ κύριε Αγγιγιόμ. Κύριο Στεμπλάς. Από την Κομισιόν θέλει να πει κάτι. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για τη συνεχιζόμενη προσοχή που δίδει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για το άσλο και συμμεριζόμαστε τα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου. Έχουμε φτάσει τώρα σε μια σταθερή λειτουργία. Έχουμε την πλήρη ικανότητα δράση του γραφείου για να μπορέσει να εξασφαλίσει την εφαρμογή του κοινού συστήματο ασύλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ο κεφαλαιόδη ρόλο του τα επόμενα χρόνια και φυσικά το γραφείο ασχολείται και με την έγκαιρη προειδοποίηση και την εφαρμογή έκτακτων μέτρων που προβλέπονται από τον κανονισμό του Δουβλίνου. <clears throat> Ευχαριστούμε λοιπόν το Κοινοβούλιο για την προσοχή που δίνει στο φορέα αυτό και την επίσκεψή του στη Μάλτα. Back to you, as head of delegation to... Κύριε Μούλτερ, ως ε, επικεφαλής αντιπροσωπείας στο ΕΑΣΟ, έχετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για το ερώτημα. Το ποιου συναντήσαμε. Είδαμε όλο το, περισσότερο προσωπικό του γραφείου ΕΑΣΟ. Μιλήσαμε με τους πρεσβευτές των κρατών μελών που εκπροσωπούνται στη Μάλτα και ακούσαμε για τις εμπειρίες τους. Τρεις υπουργούς νομίζω συναντήσαμε της τωρινής κυβέρνησης της Μάλτας. Δύο, δύο, όχι τρεις, δύο. Υπερβάλλω κατά 50%. και φυσικά και εκπροσώπους αντιπολίτευσης. Τρία σημαντικά λοιπόν άτομα σε πολιτικό επίπεδο για την Μαλτά και είχαμε στη συνέχεια μια συζήτηση όπου παρουσιάσαμε σε ένα ευρύτερο κοινό την άποψή μας, το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συζητήσαμε και με άτομα από το κοινό. Ήταν περίπου 50-60 παριστάμενοι και φυσικά μπορούσαν να θέσουν ό,τι ερωτήματα θέλανε. και συζητήσαμε και με ένα από τους ετούντες ασύλου που είχε έρθει από την Ερυθρέα και είχε ζήσει στη Λιβύη σε φρικτές συνθήκες και τώρα έχει πάρει άσυλο και θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και την επόμενη μέρα, γιατί ήταν μόνο δύο μέρες αυτή η συζήτηση, η συνάντηση, η επίσκεψη, είχαμε συζήτηση με τους ε, οι υπεύθυνου του ΕΑΣΟ που μας εξηγούσαν τι κάνουν για να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις <clears throat> και πώς, και πώς βοηθούν τους ζητούντες άσυλο και πώς κάνουν την κατάρτιση. Για το ερώτημα της κυρίας Γιλιόμ δεν νομίζω ότι κατάλαβα πολύ καλά τι εννοούσε, αλλά προς το παρόν η εντολή του ΕΑΣΟ πιστεύω ότι είναι επαρκής όπως είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν έχει φτάσει στην πλήρη του λειτουργία και αν χρειαστούν και άλλες ε, δραστηριότητες στο μέλλον. Μπορεί, αλλά δεν έχω ακούσει κάποια τέτοια... τέτοια ε, δεν καταλάβατε το ερώτημά σας κύριε Γιγιά συγγνώμη. Να είμαι πιο συγκεκριμένη για να καταλάβει ο κ. Μούλτερ. Δεν αναφερόμουν στην διεύρυνση της εντολής του ΕΑΣΟ. Έλεγα ότι μέσα στην ε, εντολή του ΕΑΣΟ υπάρχουν προφανώς τα θέματα κατεπίγουσας αντιμετώπισης που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη Μάλτα, αλλά πρέπει να υπάρχει και όλη η τακτική παρακολούθηση των θεμάτων ασύλου. Δεν πρόκειται για να διευρυνθεί λοιπόν η εντολή του ΕΑΣΟ. Δεν κατάλαβα καλά το ερώτημα. Είναι δύσκολο μετά από μια μισή μέρα να μιλήσω με κάποια αυθεντία. Για μένα νομίζω ότι το γραφείο αυτό κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του και δεν έχω κάποια αντίθετη, δεν έχω ακούσει κάποια αντίθετη άποψη. Αν υπάρχει παραμέληση των καθηκόντων του ΕΑΣΟ θα ήθελα να το ακούσω, αλλά η δική μου εντύπωση δεν υπήρξε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Εντάξει. Εντάξει, σας ευχαριστώ κύριε Μούλτερ. 12 πρέπει να τελειώσουμε, 12 και 1 είναι τώρα. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και στις 9 την πέμπτη, την επόμενη πέμπτη στις Βρυξέλλες θα έχουμε συνεδρίαση πάλι. Ευχαριστώ, γεια σας.